Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Άρχεται η συνεδρία της Υποεπιτροπής Ασφάλειας στα Πολωνικά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Σήμερα Έχουμε διερμηνία για τα τακτικά μέλη της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Το κανονικό, δηλαδή, γλωσσικό καθεστώς για την Υποεπιτροπή μας. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τη διερμηνία σε μερικές καμπύρες. Ξαναρχίζω, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν διερμηνία για τις γλώσσες των τακτικών μελών της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Μάλιστα, η συνεδρίαση μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Μην το ξεχνάτε. Περνάμε τώρα στο πρώτο σημείο, την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έγιναν κάποιες αλλαγές στις τελευταίες στιγμής. Η κυρία Αρνό, η Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, δεν μπόρεσε να έρθει, ακύρωσε την τελευταία στιγμή την ε, παρουσία της. Αποφασίσαμε λοιπόν με τη γραμματεία να καλύψουμε αυτό το κενό, αντικαθιστώντας το με ένα άλλο θέμα που έχει άμεση σχέση με το κυρίως θέμα της ε, σημερινής συνεδρίασης, το σημείο 4 δηλαδή, που προβλέπει η παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την ε, στρατηγική της ασφάλειας στην αυσιπλοεία. Μία πρωτοβουλία της Ιταλικής Προεδρίας. Θα έχουμε παρουσίαση της στρατηγικής αυτής από τρεις ε, εμπειρογνώμονες τον εκπρόσωπο της Ιταλικής Προεδρίας, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αντικατάσταση της ε, παρουσίας από τη Γενική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας αποφασίσαμε να συζητήσουμε το θέμα της ασφάλειας στη Βαλτική θάλασσα. Στις, σε μία από τις επόμενες ε, συνεδριάσεις μας, ε, όπως και σε αυτή, είπαμε ότι θα ολοκληρώσουμε την επισκόπηση της ε, κατάστασης ασφάλειας ε, σε όλες τις θάλασσες και ε, οι θαλάσσιες λεκάνες που είναι το αντικείμενο της στρατηγικής ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Για παράδειγμα, Εύξηνος Πόντος, Μεσόγειος, Θάλασσα, παρόλο που σήμερα θα ακούσουμε σχετική παρουσίαση. Θα ασχοληθούμε και με το θέμα της πειρατείας, όπως πάντα, της πειρατείας στο κέρας της Αφρικής, ή στα ύδατα γύρω από το κέρας της Αφρικής. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 3 της σημερινής διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Άιρις Ρικβέιλης, που είναι σύμβουλος άμυνας στο ΝΑΤΟ από την Λετωνία και μέλος αντιπροσωπείας της Λετωνίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Στρατηγικών Σπουδών από την Πολωνία, τον κύριο Τόμας Σατκόφσκι. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα ήθελα να εγκρίνουμε την σε διάταξη. Συμφωνείτε. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε στο σημείο 3. Παρουσίαση της κατάστασης ε, της ασφάλειας στη Βαλτική. Θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Άιρις Ρικ Βέιλις, που είναι σύμβουλος άμυνας και σύμβουλος για στρατητικά θέματα της Λετωνίας και μετά στον κύριο Σατκόφσκι. Κύριε Ρικ Βέιλις, έχετε το λόγο. Thank um, Good morning. Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στην Επιτροπή σας να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ ευρύ, πάρα πολύ περίπλοκο και δεν θα μπορέσω να χύξω όλα τα επιμέρους ζητήματα σε σχέση με τις αλλαγές όσον αφορά την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής. Θα εστιάσουμε προσοχή μας περισσότερο στα στρατιωτικά και να απαντήσουμε τυχόν ερωτήσεις. παρά τις ε, ρητορικές, τις δηλώσεις για τα όσα έχουν γίνει από πλευράς Ρωσίας φέτος αλλά και πέρσι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το ότι το Δεκέμβριο του 2007 η Ρωσία έφυγε από την ε, συνθήκη of Georgia's 2008 για τα σημαντικά στεγνώματα στην Ευρώπη. Είδαμε τι έγινε με την Ουκρανία και είδαμε τι έγινε επίσης και με την Γεωργία. Κατόπιν είχαμε ε, την ε, παρέμβαση στα εσωτερικά της Ουκρανίας και οπότε οι Ουκρανοί θέλησαν να έχουν πιο στενούς δεσμούς τότε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι ξεπλάγησαν όταν ε, κατεληφθεί η Κρυμαία τον Μάρτιο του 2014 και είχαμε και την εξέγερση στην Ανατολική Ουκρανία και κατόπιν την διείσδυση του Ρωσικού στρατού το 2014 πάντα, οπότε θα πρέπει να δούμε τα όσα έγιναν στην Ουκρανία στο ευρύτερο πλαίσιο όσων έγιναν στην περιοχή. Όλα αυτά είχαν σημασία μεγάλη και για την ασφάλεια στη Βαλτική. Τα τελευταία χρόνια εκεί είδαμε μια αύξηση στις εθνικές δραστηριότητες κοντά στα σύνορα των βαλτικών χωρών της Πολωνίας και της ε, περιοχής γενικότερα. Όλο ένα και περισσότερο αυξάνουν οι δαπάνες και εξυγωνισμός του στρατού της Ρωσίας, το σχετικό πρόγραμμα που κοστίζει πολλά εκατομμύρια. Οπότε θα σας πω με λίγα λόγια τι ότι ανέπτυξε στην περιοχή της Βαλτικής η Ρωσία. Ενίσχυσαν τις δυνάμεις στις όμορες χώρες, τακτικά κάνουν στρατηγικές ε, ασκήσεις και ενίσχυσαν τις ε, δυνατότητές τους για να μπορούν να χτυπήσουν μακριά. Επίσης αυτό έγινε και όσον αφορά την παρακολούθηση των δυνατοτήτων των γειτονικών χωρών για να τους ανασχέσουν ευθές οι χώρες. Είδαμε τι έγινε επίσης σε Ουκρανία και Γεωργία. Πέμπτον, είχαμε επίσης αύξηση της πίεσης πλευράς διπλωματίας και υπηρεσιών πληροφοριών εκ των ε, μέσω της ενεργικής πολιτικής πιέζουν τις όμορες χώρες και είχαμε αυτές τις έξι Οπότε ανασταθούμε στα θέματα καθαρά ασφάλειας, δηλαδή στα πρώτα τρία από πούμε και κάποια στοιχεία. Επιδεικνύει τη δυναμή της η Ρωσία από το Σεπτέμβριο του 2009 και η Λευκορωσία με τη Ρωσία κάναν την άσκηση ΖΑΠΑ του 2009. Και οι ασκήσεις αυτές ε, ε, ήταν γυμνάσια σε σχέση με επίθεση στο ΝΑΤΟ είσαι στι ε, βαλτικέ χώρες, 12.500 στρατιώτε, 6.000 ήταν από τη Ρωσία, 40 αεροπλάνα και 200 άλλα στρατιωτικά οχήματα. Οπότε βλέπουμε τι έγινε το 2009-2010 ανακοίνωσαν, ανακοίνωσαν μαζικό εξοπλισμό 720 δις δολαρίων, 70% του υλικού του θετικού θα αντικατασταθεί και επίσης ο προϋπολογισμός υπερδιπλασιάστηκε από το 2007. Το Σεπτέμβριο του 2013 η Ρωσία και η Λευκορωσία κάναν την άσκηση Ζάπα το 2013 και επίσημα αυτό ονομαζόταν ως αντιτρομοκρατική άσκηση. Και αυτό ήταν μια άσκηση επίθεσης στις ε, γειτονικέ χώρες. Και το ΖΑΠ 2013 είχε 12.900 στρατιώτες και ε, περισσότερο ε, από τη Ρωσία 70 τεθωρακισμένα και ε, συμμετέσχε και η Λευκορωσία όπως είπαμε αλλά και σκάφη από τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Άλλα στοιχεία ήταν τα επίσημα και άλλα ήταν τα πραγματικά στοιχεία του το, το, στρατού που συμμετέσχε. Και εκτός από τους βασικούς στόχους, επίσης, ε, συμμετέσχε και το Υπουργείο Μεταφορών και μετακίνησαν πάρα πολύ υλικό σε μεγάλες ε, αποστάσεις και στόχος ήταν είναι τα δυτικά σύνορα και είπαν και επίσης στο Καλίνγκρατ πήγαν πάρα πολλά πυραυλικά συστήματα σύμφωνα με στοιχεία του ΝΑΤΟ. και μπορούν να χτυπήσουν στόχους τώρα σε Πολωνία, Γερμανία και σε βαλτικές χώρες. Το Δεκέμβριο του 2013 η η Ρωσία ξανά άνοιξε μια βάση 32 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Λετωνίας και κάποια μοίρα αεροπορίας με κάποια βάση τέλος πάντων την ενεργοποίησαν πολλά σκάφη ήταν εκεί και ελικόπτερα αυτή η βάση Όστρο είναι πάρα πολύ κοντά στις πρωτεύουσες της Βαλτικής, αλλά και στη Φιλανδία. Από εκεί μπορεί κανείς να χτυπήσει ή μπορεί να φτάσει τέλο πάντων στην, ε, στην Το 2014 ε, απήγαγαν κάποιον Λετωνό ο οποίο μετάφραγε στη Μόσχα και, και επίσης λιθουανικό σκάφος ε, ε, κατασχέθηκε από τις Ρωσικέ αρχές και επίσης υπήρξαν και παρενοχλήσεις φιλανδικών ε, σκαφών και κάποια υποβρύχια έφτασαν μέχρι την Σουηδία, υποβρύχια ρωσικά, τον, από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 αυξήθηκε η στρατιωτική δραστηριότητα. Πολύ κοντά στην Λετωνία. Εννέα μήνες, κατά το 2014, είχαμε περίπου 170 περιπτώσεις που είχαμε υπερπτήσεις ε, αεροπλάνων αλλά και ναυτική δραστηριότητα. Όλα αυτά δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Και σε σχέση με το ας πούμε, που είχαμε μόνο τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις. Παραβίαση του Σουηδικού ε, χώρου 23 φορές και 17 ένα άλλο μήνα και στις περισσότερες αυτές τις περιπτώσεις τα ρωσικά αεροπλάνα αλλά και σκάφη δεν παραβίασαν τα διεθνή σύνορα αλλά δεν ανταποκρίθηκαν το κάλεσμα το θεμητό των βαλτικών ε, χωρών να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Επίσης, παραβίαση του φιλανδικού ενεργείου χώρου Μάιο, Αύγουστο και Οκτώβριο. Στις 21 Οκτωβρίου για έκτη φορά παραβίασαν τον ιστονικό ενέργειο χώρο. Τέλειο Οκτωβρίου είχαμε διάφορες υπερπτήσει ε, στην Ευρώπη μέχρι και την Πορτογαλία και επίσης στη Βαλτική αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης ε, όσον αφορά την Βαλτική και δραστηριότητα των Ρώσων βλέπουμε ότι το Μάιο του 2014 το ρωσικό ναυτικό έκανε κάποιες ασκήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λιθουανίας και έτσι τα λιθουανικά πλοία δεν μπόρεσαν να ε, πάνε εκεί που πηγαίνανε προηγουμένως και στην Λετωνία το ίδιο με αναγνωριστικά, με κορβέτες και με υποβρύχια. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο να προκαλέσουν και να δοκιμάσουν την ε, δυνατότητα αντίδρασης των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Επίσης, κάνουν έτσι επίδειξη δύναμης. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό με τα πολεμικά ή τέλος πάντων μετά τον ψυχρό πόλεμο. Τώρα που συζητούμε συνεχίζουν αυτές τις δεν πρόκειται όμως για μεμονωμένα περιστατικά, ούτε πρόκειται για κάποιες συμπτώσεις σε χώρο και χρόνο. Είναι κάτι το γίνεται επίτηδες και ε, οπωσδήποτε πρόκειται για μια μακρόπνοη πολιτική αντιπαράθεσης με τους γείτονες στη Βαλτική και σε άλλες περιοχές. Σαν αποτέλεσμα τούτου είδαμε τη συζήτηση έγινε, τι αποφάσεις ελήφθησαν όσον αφορά ε, το, τις δαπάνες τις Είδαμε τι έγινε σε Σουηδία και Φιλανδία για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Είδαμε επίσης ε, ε, την αυξημένη συνεργασία στην Βαλτική και επίσης ασκήσεις ε, των νατοικών δυνάμεων στην περιοχή αυτή. Thank you. Thank you. Um, um, yes, um, and in practical um, terms they cannot be even... Οπότε δεν είναι δυνατόν καμία δραστηριότητα να συγκριθεί με τη ρωσική δραστηριότητα στην περιοχή. Αν το δούμε ευρύτερα το θέμα αλλά και στατικικά, αυτή η δραστηριότητα θέλει να αποδομήσει την κατάσταση της ασφάλειας μετά τον ψυχρό και επίσης δημιουργούνται και κάποιες ε, αμφιβολίες ε, έτσι για την αρχιτεκτονική της ασφάλειας στην Ευρώπη μετά τον ε, πόλεμο όπου το βασικό θεμέλιο, η βασική αρχή ήταν το απαραβίαστο των συνόρων. Τι μπορεί να γίνει. βεβαίως και υπάρχουν κάποιες μελέτες, κάποιες ιδέες για το τι πρέπει να κάνει το κάθε κράτος για την άμυνα και τις στρατιωτικές δυνατότητες και, και η δική μου κυβέρνηση αλλά και το Κοινοβούλιο της Λετωνίας αποφάσισε βαθμία να αυξηθεί μέχρι το 2020 η δαπάνη για την άμυνα ε, και να φτάσει το 2% του ΑΕΠ μας. Έχουμε κάποιους επίσης λογικούς ε, στόχους που θα πρέπει να σας ε, εξηγήσω. Πρώτα πρώτο πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει αυξηθεί σημαντικά. Η κυρία έχει γνώμη τώρα έχει εξελιχθεί από τότε που υπήρχε κάποια διαφοροποίηση για το ότι ήταν κακό το ΝΑΤΟ καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ ουσιαστικά αποτελούν ε, ενιαία και αδιαχώριστα εχθρό αντίπαλο. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό, θα μπορεί να γίνει τώρα συντονισμός και να πάμε σε μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα αυτών των δύο οργανισμών. Οπότε και θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό το ΝΑΤΟ αν θέλουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό. Οπότε θα πρέπει να έχουμε περισσότερο προσωπικό και στις δύο οργανισμούς και οπότε θα πρέπει να διευρυνθεί η δραστηριότητα αυτού του προσωπικού. Συνεργασία και επίσης να ακούγεται η φωνή, να ακούγεται με μία φωνή η άποψη αυτών των οργανισμών. Τα βασικά κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι απλώς 6 χιλιόμετρα μακριά από το ΝΑΤΟ και έχουμε 28 μέλη ε, της αντιπροσωπείας που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και δύο οργανισμοί Τώρα δεν έχουν ε, ε, ενία τοποθέτηση. Στην Ουαλία έγινε μια σύνοδος και είπαμε ότι εκεί υπάρχει μια διαφορά. Τώρα πια σχέση με πριν μετά τόσα έγινε στην Ουκρανία. Εμείς σου πω πώς ε, ερμηνεύουμε τα πράγματα μετά από την τελευταία Ευρωπαϊκή Σύνοδο πριν από δύο μέρες. Είπαμε ότι από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαπιστώθηκε ε, ότι υπάρχει βούληση συζήτηση για το τι έγινε στην Ουκρανία όμως οι απειλές είναι περισσότερες και θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν όλες αλλά θα πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση περιφερειακές ε, απειλές σε σχέση με άλλες απειλές αυτές που μπορούν να έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις και είναι και πυρηνικού χαρακτήρα. Χρειάζεται μόνο μια στρατηγική, χρειάζεται ε, να λάβουμε υπόψη το πόσε ε, απόψεις έχουν διατυπωθεί και έχουμε μια έκθεση από την υπάτη εκπρόσωπο το οποίο θα πρέπει να προετοιμάσει ένα συμβούλιο το 2015 τον Ιούνιο. Θα γίνει αυτό στην Ρήγα, οπότε εκεί μπορούμε να συμφωνήσουμε για το πώς θα αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας. Άλλο θέμα είναι η ασφάλεια των συνόρων. Επί μακρόν εστιάζουμε προσοχή μας στην ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων σε σχέση με την λαθρομετανάστευση και το λαθρεμπόριο ε, υπηρεσιών και εμπορευμάτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε προοδεύσει εκεί σε αυτά τα σημεία και πιστεύουμε ότι η Λετωνία και άλλα κρατημέλη έχουν αναπτύξει πάρα πολλά διαφορετικά μέτρα, εφαρμόσιμα επιτόπου, καλό συντονισμό και ανταλλαγή πληρονομιών. Επίσης, όσον αφορά νόμες δραστηριότητες για τα θαλάσσια σύνορα. Όμως, δυστυχώς, αυτά που κάνει η Ρωσία υπονομεύουν την ε, υγιή συνεργασία με την Ρωσία όσον αφορά την ασφάλεια των σύνορων, κάτι το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια. Και ε, ε, το ότι δεν συμμορφώνεται η Ρωσία με το διεθνές δίκαιο ε, γι' αυτό συνεχίζεται, αυτό φέρνει μεγάλη αβεβαιότητα και αυτό πλήσει επίσης την συνεργασία. Επίσης, σε σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα, θα πρέπει να πούμε το ότι η ασφάλεια των συνόρων ε, έχει σχέση με διάφορες δραστηριότητε και την λαθρομετανάστευση, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε αυτή η ασφάλεια. Το είδαμε αυτό από τα όσα κάνει η Ρωσία στην ε, Ουκρανία, αλλά και στην Εστονία. Οπότε η ασφάλεια των συνόρων είναι διαφορετικό περιεχόμενο πέραν του παραδοσιακού. Άρα τώρα θα πρέπει να έχουμε με ένα μεγάλο φάσμα ε, μέσων και μέτρων. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε αυτές τις υβριδικές απειλές, τι επιπτώσεις έχουν για τους ε, πολίτες μας, γιατί αυτού του είδους ο υβριδικός πόλεμος μπορεί να έχει πολλές μορφές σε σχέση με τις συμβατικές ε, επιχειρήσεις, ε, τον ανταρτοπόλεμο, ε, κυβερνοπόλεμο, άρα θα πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε την ασφάλεια των συνόρων μας, άρα στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τη συλλογή πληροφοριών για τις ε, δραστηριότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των δορυφόρων της. Και από ανοιχτέ πηγές και από πλήσεις πληροφοριών και να είμαστε περισσότερο ε, να έχουμε δυνάμεις ασφαλείας που είναι πιο καλά προετοιμασμένες για να μπορούν να ανταποκριθούν αν χρειαστεί. Επίσης, από τη φύση του αυτός ο ευρωδικός πόλεμος είναι τέτοιος που δείχνει, είναι κάτι σαν κοινωνική αναταραχή κάτι το οποίο θεωρούμε στις κοινωνίες μας ότι είναι κάτι το θεμητό και ότι είναι συμβάν, είναι εκδηλώσεις τέλος πάντων της δημοκρατίας. Επίσης θα πρέπει να σας τονίσω το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε συνέργεια του, του, του θεωρητικού τομέα με τον πολιτικό, ε, εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια τώρα δεν, δεν έχει κάποια διαφορά. Έχουμε τις πανδημίες, έχουμε τον υβριδικό πόλεμο, όλα αυτά φέραν αυτή την αλλαγή και σας ε, υπενθυμίζω ότι όλα τα χρωτοφυλάκια των επιτρόπων έχουν μέσα και θέματα ε, ασφάλειας, που θα πρέπει να υπάρχει και ένας αντιπρόεδρος στην επιτροπή για να συντονίζει σε σχέση με όλα αυτά. Οπότε... Η Λετωνία συνεχίζει να είναι υπέρ ισχυρών δεσμών με τον ΝΑΤΟ και ενίσχυση της συμπληρωματικότητα των επιχειρήσεων που θα πρέπει να αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης των ικανοτήτων μας σε μια κατάσταση διαχείρισης των παγκόσμιων κρίσεων. Επίσης θα πρέπει να συσφίξουμε τις σχέσεις με τους πιο σημαντικούς συμμάχους μας, Ηνωμένε Πολιτείε, Καναδά, Νορβηγία και Τουρκία. Ένα άλλο σημείο είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια αναπτύσσαμε περιφερειακή συνεργασία και σχετική εμπειρογνωσία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Είχαμε με τη Βαλτική Βίσεγκραντ ε, και άλλους σχηματισμούς θα πρέπει να τις συνδυάσουμε με πρωτοβουλίες ε, των συνδυασμένων δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ώστε όλα τα κράτη-μέλη να βρουν ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος συμμετοχής σε τέτοιες ε, συνεργασίες και να ενισχύσουν την ασφάλειά τους. Επίσης, θα πρέπει να κρατήσουμε την επαγρύπνησή μας σε σχέση με την προπαγάνδα που κάνει η Ρωσία και εντός και εκτός. Είναι πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα και έχει νομικά, πολιτικά στοιχεία και είναι και θέματα αξιών. Δεν πρόκειται να εντρυφήσω σε λεπτομέρειες. Πάντως το θέμα της πληροφορίας και της χειραγώγησης των, της πληροφορίας είναι βασικό στοιχείο του πολέμου και η πρόσβαση σε ε, πηγές πληροφόρησης ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, ας μην ξεχνούμε και την ικανότητα που έχει πλήση εγκεφάλου, που στόχο έχει την αποδυνάμωση της ενότητας και τη διάβρωση της γενικής επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε πια την πολυτέλεια της ασφάλειας και της ειρήνης όπως νομίζαμε ότι θα είχαμε μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης γιατί έχουμε πόλεμο ουσιαστικά 2.000 χιλιόμετρα από, την, από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι τόσο μακριά λοιπόν όπως βλέπετε. Επίσης ε, η ασφάλεια της Βαλτικής θάλασσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εμείνουμε στην εσωμάτωση ε, και στην ολοκλήρωση του ΝΑΤΟ γιατί η ασφάλειά μας είναι μια διαδικασία αν το γίγνεσθε και επίση θα πρέπει να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση τη σταθερότητα και τη ασφάλεια και στη γειτονία μα και να αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνού δικαίου. Έτσι θα πρέπει να αποτρέψουμε όσους θέλουν να μας αποσπάσουν την προσοχή από τις θεμελιώδεις αρχές και ελευθερίες μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρικ Και παρακαλώ παραμείνετε για να δώσετε απαντήσεις και να λάβετε μέρος στη συζήτηση. Ο λόγος τώρα στον κύριο Τόμας Σατκόφσκι. Mr. Rukvelis gave, a very interesting overview of Russian activity in, the, in the region. Therefore, I will move on a little bit, starting off with a broader depiction of the, of the, of the meaning. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω με μια ευρύτερη εικόνα της ε, γεωπολιτικής ε, διάστασης και μετά θα περιγράψω την, ε, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης της Βαλτικής και να αναφέρω κάποια στρατιωτικά σενάρια και σενάρια ασφαλείας και τέλος θα αναφέρω το τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη δυνατοτήτων στην περιοχή. Ξεκινώντας με την Βαλτική και το Καλίνιγκραντ. Όσο η Ρωσία δεν μπορεί να ελεγχεί τον κύριο όγκο της ε, Ουκρανικής ε, επικράτειας, ε, ούτε της Λευκορωσίας, τουλάχιστον καιρό ειρήνης, η αντιπαράθεση με την ευρύτερη δύση περιορίζεται στην Βαλτική και στην ε, υποαρκτική περιοχή. Και συνδέονται αυτές οι περιοχές ε, και η μία επηρεάζει την ε, άλλη. Όπως πάρα πολλοί ε, Βρετανοί έχουν επισημάνει, η πρόσβαση στην ε, Βαλτική έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καθώς επίσης ε, και η περιοχή μεταξύ Βαλτικής και Μαύρης Θάλασσας. Το Καλίνιγκραντ θεωρείται ένα σημείο προβληματικό το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο των βαλτικών ε, κρατών. Ιστορικά η Βαλτική ήταν ε, μεγάλη σημασία για διάφορους λόγους. Οικονομικά πρώτα απ' όλα ήταν πηγή πρώτων υλών που έφευγαν προς τις ε, δυτικές χώρες. Ε, ξυλία, σίδηρο, χαλκό κτλ. Σήμερα έχει επίσης μεγάλη εμπορική σημασία, όπως δείχνουν οι έρευνες. Γύρω στα 100.000 ε, σκάφη το χρόνο διασχίζουν την ε, Βαλτική. Οι πρώτες ε, ύλες και η εξαγωγή τους από τον Πυθμένα έχει ενταθεί. Υπάρχει και η γνωστή περίπτωση του αγωγού Nord Stream, ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ρωσία στη Γερμανία και ο οποίος λειτουργεί εξάρτηση βεβαίως των χωρών που βρέχονται από την Βαλτική, από τους ε, θαλασσίους διάβλους επηρεάζει την ευημερία τους. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η Βαλτική δεν ήταν ε, ένα θέατρο μεγάλης ε, σημασίας για τη στρατηγική της Δυτικής Συμμαχίας, όμως ο έλεγχος των στενών της Δανίας είχε μεγάλη σημασία γιατί εάν ε, τα καταλάμβανε αυτά η Σοβιετική Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση προβολής ισχύω του Σοβιετικού Ναυτικού στην ανοιχτή θάλασσα και βεβαίως να περιπλέξει την κατάσταση για τις ενισχύσεις ε, που θα έρχονταν ε, στη Δυτική Ευρώπη. Η Βαλτική είχε επίσης μεγάλη σημασία από πλευράς ε, ναυπηγείων και οι Σοβιετικοί είχαν ε, τον κύριο όγκο των ναυπηγείων τους εκεί. Επίσης η εκπαίδευση του Σοβιετικού και του Γερμανικού ναυτικού ε, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε εκεί κατά κύριο λόγο. Τώρα, να περάσουμε στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της ε, Βαλτικής. Η Βαλτική έχει μήκος 700 ναυτικά μίλια και πλάτος ε, μεταξύ 100 και 200 ναυτικών μιλίων. Ε, έχει δηλαδή ένα μακρόστενο σχήμα κάτι το οποίο έχει στρατιωτικές επιπτώσεις τις οποίες θα αναφέρω στη συνέχεια. Στρατηγικά σημεία, όπως ανέφερα, τα στενά της Δανίας ε, που έχουν τεράστια σημασία. Όποιος, τα ελέγχει ε, μπορεί να επηρεάσει την ευημερία των άλλων κρατών που βρέχονται από τη Βαλτική. Οι άλλε έξοδοι είναι... Ε, του Κιέλου και βεβαίως και ο διάβλος ε, της θάλασσας του Μπάρεντς ε, που κατασκευάστηκε επί Σοβιετικής Ένωσης που μπορούν εύκολα να μπλοκαριστούν σε περίοδο εχθοπράξεων. Υπάρχει επίσης ε, και η στενή έξοδος του κόλπου της ε, Φιλανδίας ε, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και βεβαίως αυτό φαίνεται από το ότι μπορούσαν οι Γερμανοί να μπλοκάρουν την έξοδο κατά τη διάρκεια του πολέμου με μερικές νάρκες που έβαλαν στον φιλανδικό κόλπο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Βαλτικής είναι ο μεγάλος αριθμός νησιών που έχει μεγάλη σημασία. Αναφέρω εδώ πέρα παραδείγματος χάρη το σουηδικό νησί Γκότλαντ που είναι στη μέση περίπου της ε, Βαλτικής και δίνει στους ε, Σουηδούς την δυνατότητα να ελέγχουν πλήρως τις κινήσεις των πλοίων. Η σημασία αυτή βεβαίω αποκαλύφθηκε και τονίστηκε και πρόσφατα καθώς και ο κίνδυνος εισβολής που υπάρχει και έχει τονιστεί ακριβώς. Τα φινλανδικά νησιά ελέγχουν ε, την είσοδο στον κόλπο της ε, Βυθνίας ε, και είχαν επίσης χρησιμοποιηθεί και σε άλλες σύγκρουσεις στο παρελθόν. Όσον αφορά τα υπόλοιπα γεωφυσικά χαρακτηριστικά είναι ρηχή θάλασσα η Βαλτική με μέγιστο βάθος 459 μέτρα η ε, περιεκτικότητα σε αλάτι είναι σχετικά χαμηλή γιατί είναι χαμηλές θερμοκρασίες και χαμηλή η εξάτμιση επίσης είναι ταραχώδης θάλασσα τι σημαίνουν τώρα αυτά για την ε, στρατιωτική ε, διάσταση λόγω ακριβώς ε, του μακρόστενου αυτού σχήματος ε, που ανέφερα μεγάλο ρόλο θα παίξει, θα παίξει και η αεροπορία και η επάκτη άμυνα, ο ναρκοπόλεμος και ο πόλεμος υποβρυχίων. Όσον αφορά λοιπόν τα τελευταία αυτά, η Βαλτική, παρά το ότι θα περίμενε κανείς, είναι πάρα πολύ καλό περιβάλλον για υποβρύχια και οι ειδικοί λένε πως είναι τέσσερις φορές πιο δύσκολο να εντοπιστεί ένα υποβρύχιο στη Βαλτική από ότι παραδείγματος χάρη στη Βόρεια Θάλασσα. Τα γεωγραφικά αυτά χαρακτηριστικά σημαίνουν πως στην περίπτωση εχθροπραξιών μεγάλης έντασης, η Βαλτική θα γίνει μια απαγορευμένη ζώνη ή νεκρή ζώνη και για τους δύο πιθανούς αντιπάλους. Αυτό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση πρώτα απ' όλα για τις βαλτικές χώρες και τις πιθανές ενισχύσεις που θα έρθουν. και το Καλίνιγκραντ ε, ακριβώς ε, δημιουργεί πρόβλημα γιατί θα έχουν μεγάλη σημασία οι χερσαίες ε, γραμμές επικοινωνίας και το Καλίνιγκραντ μπορεί να εμποδίσει ακριβώς τις ενισχύσεις. το Καλίνιγκραντ ε, μπορεί να γίνει ακριβώς ένα αγκάθι στα μετόπισθεν με βάση και βάση για πυρευλικά διαρροπορικά στήματα Ισκαντέρ και για Χόντ. Αναφέρθηκα στην στρατιωτική διάσταση και ίσως αναρωτηθείτε τι σημασία έχει πλέον μιας που οι Ρώσοι έδειξαν προτίμηση σε μη συμβατικά και παραδοσιακά μέσα για την αύξηση της επιρροής τους, ενεργειακούς εκβιασμούς, ε, οικονομικό πόλεμο κτλ. Και τα μικρά πράσινα ανθρωπάκια που είδαμε στην Ουκρανία. Αλλά θα μιλάμε για το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα. Οι Ρώσοι δηλώνουν ανοιχτά ότι αν αποτύχουν τα πιο μαλακά ήπια μέσα θα προσφύγουν σε ε, πιο δυναμικά και η σύγκρουση του Ντομπάς το απέδειξε. Όσον αφορά λοιπόν τις προθέσεις της Ρωσίας που μπορεί κάποιος ε, για τις οποίες μπορεί κάποιος να αμφιβάλλει είναι δύσκολο να κρίνουμε εάν πρόκειται για κάποιον ε, εκβιασμό που στόχο έχει την εδραίωση της εξουσίας ε, σε σχέση με το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας ή αν είναι μια προσπάθεια να ανακαταληφθούν περιοχές που ήταν κάποτε υπορωσική επιρροή ή απλά να αλλάξουν οι κανόνες του γεωπολιτικού παιχνιδιού πριν είτε ε, πρώτον η Ρωσία λόγω της ενεργειακής επανάστασης χάσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί πλέον τον στρατό της ή β εκλεγεί ένας πιο αποφασιστικός Αμερικανός πρόεδρος. Τέλος η σύγκρουση που α, ε, πιθανώς ε, θα έχει και οικονομική και πολιτική ε, διάσταση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αντίληψη που υπάρχει για τη στρατιωτική ισορροπία. Γι' αυτό έχει σημασία και η στρατιωτική ισορροπία. Και για να επανέλθω στην στρατιωτική ισορροπία, ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ρικβέλης ανέφερε το υβριδικό σενάριο. Όμως, το να γνωρίζουμε, γνωρίζοντας ε, τις ε, ε, έννοιες του ρωσικού στρατιωτικού δόγματος, αν αποτύχουν αυτά τα υβριδικά μέσα, η Ρωσία θα προσφύγει σε πόλεμο. Επίσης μπορεί να υπάρξει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία ίσως επιτεθεί στην Πολωνία στόχο να συντρίψει όλη την περιοχή γιατί εάν ε, καταβληθεί η άμυνα της ε, Πολωνίας πλέον οι υπόλοιπες χώρες, οι βαλτικές έχουν τελειώσει το... για το τι μπορεί λοιπόν να γίνει πρέπει να έχουμε κατά νου τις δυνατότητες ε, άρνησης ε, περιοχής ε, και άρνησης πρόσβασης που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι δυνατότητες αυτές αναπτύχθηκαν για να ακυρώσουν τις δυτικές δυνατότητες προβολής ισχύω. Και εδώ πέρα αναφέρομαι σε εξελιγμένες δυνατότητες αεράμνας S300, S400 για χόντ, βλήματα κατά και τα βαλιστικά βλήματα Ισκαντέρ και βλήματα πλεύσης επίσης. Πυροβολικό και βέβαιως ε, συστήματα ραδιοηλεκτρονικά. Επίσης υπάρχουν ε, επιχειρησιακές ε, μονάδες ελιγμών σχεδιασμένες για διείσδυση, για βαθία διείσδυση και με μεγάλη ευελιξία. Και όσον αφορά λοιπόν το υβριδικό λεγόμενο σενάριο, δεν έχει, δεν έχει εκεί πέρα τόσο μεγάλη σημασία η ποιες είναι οι δυνατότητες και οι αριθμοί, αλλά η πολιτική βούληση. Δηλαδή μπροστά σε μια τέτοια απειλή ο αντίπαλος είτε θα ε, υποχωρήσει είτε θα καταφύγει σε παραδοσιακό συμβατικό πόλεμο. Και εδώ πέρα ακριβώ χρειάζεται μια αλλαγή ε, λογικής και παραδείγματος. Τα τελευταία 20 χρόνια τονίζουμε την ποιότητα αντί για την ποσότητα, την προβολή ισχύω καθώς επίσης ε, και τον αντιαντάρτικο αγώνα αντί για τις ε, κλασικές ε, δυνατότητες. Στην περίπτωση λοιπόν της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αλλάξει η λογική. Οι χώρες της περιοχής πρέπει να σκεφτούν περισσότερο τις δυνάμεις τοπικής άμυνας και την ισχύ πυρός. Υπάρχει άλλη μια διάσταση του πολέμου που είναι πάρα πολύ σημαντική είναι το έλλειμμα πυρηνικής αποτροπής που προβληματίζει στην περιοχή. Κατά βάση, αν δούμε την ισορροπία δυνάμεων, υπάρχει μια στρατηγική ισοδυναμία ΙΠΑ και ε, Ρωσίας ε, ε, και υπάρχει βεβαίως και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, αλλά στις, ε, στα τακτικά πυρηνικά όπλα υπάρχει ένα κενό. Η Ρωσία έχει γύρω στις 3.000 ε, τακτικές πυρηνικές κεφαλές και έχει και εξελιγμένα συστήματα μεταφοράς τους. Επιπλέον ε, επεξεργάζεται κάποιες νέες ιδέες όπως περιορισμένη χρήση αυτών των όπλων σε ένα στρατιωτικό σενάριο. Και αυτό το οποίο κάνει αυτά τα σενάρια πιο ρεαλιστικά είναι το γεγονός πως η Ρωσία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το μέγεθος αυτών των κεφαλών και να τα βάλει σε νέους φορείς όπως ε, παραδείγματος χάρη πυροβόλα κολίτσια ή βλήματα Ισκαντέρ. Ένα άλλο θέμα είναι η παραβίαση της ε, συνθήκης ε, για τις ε, πυρηνικές δυνάμεις και αυτό σημαίνει, όπως επιβεβαίωσαν οι είπα, και αυτό σημαίνει πως η Ρωσία θα μπορεί να κάνει έναν περιορισμένο πυρηνικό πόλεμο κατά ευρωπαϊκών χωρών. Θα τα θυμάστε αυτά με την ε, στάθμευση βλημάτων ε, ε, πλεύσης στη δεκαετία του 80 στην Ευρώπη. Αλλά όσον αφορά τώρα την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας η ιδέα αυτή των σχηματισμών μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσφέρει τίποτα σε αυτό το σενάριο και πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο. Επίσης, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για να διασφαλιστεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Σουηδίας, Φιλανδίας και χωρών του ΝΑΤΟ για πόλεμο συμβατικό και υψηλής έντασης. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σατκόφσκι. Και τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Ακούσαμε από τους δύο καλεσμένους μια γενική επισκόπηση της κατάστασης και ποιες ε, προκλήσεις εκκρεμούν στην περιοχή την ευρύτερη περιοχή, γιατί έχουμε και την περιοχή Intermarium, ανάμεσα στις δύο θάλασσες, της Βαλτικής και της Μαύρης θάλασσας. Πολύ σημαντικό και αυτό το σημείο. Και η μνήα του πολέμου της πληροφορίας είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης ε, η πιθανότητα κάποιων μέτρων υβριδικού πολέμου. Και αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ εντυπωσιακά στοιχεία, γιατί τέτοιου είδους δραστηριότητε αυτή τη στιγμή και επιχειρήσεις παρατηρούμε σε όλες τις ε, χώρες της περιοχής. Η παρουσίαση του κυρίου Σατκόφσκι αφορούσε περισσότερο υποθετικά μελλοντικά σενάρια και δυστυχώς όλα αυτά τα σενάρια όσο υποθετικά και αν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη Μπορούμε τώρα να περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριος Στετίνα ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικός. Πρόσφατα ήμουνα στο Χονγκ και συζήτησα με κάποιους ντόπιου για τη Ρωσία και τους Ρώσους και μου είπαν «Α, είναι αυτή η αιμοβόρα φιλή που κατοικεί στο βορρά. Αυτή δεν είναι η Ρώση». Και μετά τις παρουσιάσεις των κυρίων Ρικβέλης και Σατκόφσκι πραγματικά θορυβήθηκα γιατί είναι πολύ ανησυχητικά αυτά που ακούσαμε. Τι γίνεται με το θύλακα του Καλινιγκράτ. Δεν αναφερθήκατε εκτενώς στο σημείο αυτό. Ποια είναι η στρατιωτική παρουσία στο Καλίνιγκρατ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζέμκε. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμότατα τους δύο καλεσμένους μας, όχι μόνο για τις πληροφορίες και την ποσότητα των πληροφοριών, αλλά κυρίως για την ποιότητα. Είναι δεύτερη φορά που είμαι μέλος της ε, υποεπιτροπής και πολύ συχνά, δυστυχώς, έχουμε πολύ γενικές και αόριστες πληροφορίες. Τόσο ειδικέ ε, και ποιοτικέ πληροφορίες ε, δεν είχαμε. Πολύ σπάνια. Συνήθως ακούμε ότι διαβάζουμε και στις εφημερίδες. Αλλά εσείς οι δύο πραγματικά αντιμετωπίσατε με πολύ σοβαρό τρόπο την Επιτροπή και μας ε, διαβιβάσετε πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και σας είμαι ευγνώμων γι' αυτό, γιατί πολύ συχνά, δυστυχώς, τα μέλη της ε, Επιτροπής αυτής ε, δεν τη χάνουν τις μεταχείρισεις που αξίζουν συνήθως οι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πάντως που εσείς ε, δεν υιοθετήσατε τέτοια συμπεριφορά και μας αντιμετωπίσατε με τη δέωση σοβαρότητα και μας δώσατε ποιοτικέ πληροφορίες. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να διαχωρίσουμε τις δύο σφαίρες δραστηριοτήτων της Ρωσίας. Και δεν μιλώ για τα γεωπολιτικά, περισσότερο για τα αποτελέσματα. Η πρώτη σφαίρα δραστηριοτήτων είναι οι προκλητικές δραστηριότητες, η επίδειξη δυνάμεως που κάνει η Ρωσία και η δοκιμασία των, α, της αντιεροπορικής άμυνας ή της δυνατότητας αναχέτησης των α, γειτονικών χωρών. Η δεύτερη σφαίρα δραστηριοτήτων, η δεύτερη κατηγορία δεν είναι μόνο προκλητικές ενέργειες, ε, αλλά η κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το σχόλιο μου αφορά περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία, τη δεύτερη σφαίρα δραστηριοτήτων, γιατί για κάθε κατηγορία οι αντιδράσεις μας θα πρέπει να είναι διαφορετικές. Έχω λοιπόν ερώτηση. Ποιες είναι οι πιθανές μας αντιδράσεις σε περίπτωση που παραβιάζεται κατάφορα το διεθνές δίκαιο από τη Ρωσία. Για παράδειγμα, όταν παραβιάζονται τα χωρικά ύδατα μιας χώρας ή όταν παραβιάζεται ο εναέριος χώρος μιας χώρας. Γιατί άλλο να πετάει κανείς στα όρια του εναέριου χώρου και να ε, προκαλεί και άλλο να παραβιάζει ενεργά τον εναέριο χώρο μιας κυρίαρχης χώρας, γιατί είναι διαφορετικές οι διαδραστηριότητες. Πόσες φορές θα δεχτούμε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και όχι, δεν μιλώ για απλές προκλήσεις, παραβίαση χωρίς να αντιδρούμε. Πόσες φορές θα δεχτούμε τέτοιες παραβιάσεις μένοντας με τα χέρια σταυρωμένα και τι θα πρέπει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν σε περίπτωση κατάφορης παραβίασης των αρχών του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Βανόρντεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους δύο προσκεκλημένους μας για τις πολύ μεστές και άρτιες παρουσιάσεις τους. Όπως συνήθως σε τέτοιες συζητήσεις διαπιστώνουμε πόσο ασήμαντη είναι η στρατιωτική ε, δύναμη και το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Και είναι διπλά ανησυχητική αυτή η κατάσταση. Γιατί όχι μόνο προσπαθούμε να διαμορφώσουμε το στρατιωτικό μας δυναμικό ξεχωριστά από το ΝΑΤΟ, αλλά η ίδια η Ρωσία προσπαθεί να διχάσει τη Δύση, αξιοποιώντας ακριβώς τις διαφορές ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακούσαμε το πρωί τη διαφορετική φρασιολογία που χρησιμοποιούν και τη διαφορετική ρητορική που χρησιμοποιούν οι δύο οργανισμοί, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις σχέσεις τους με τη Ρωσία. Βέβαια φαίνεται ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πολύ πιο σοβαρά το ΝΑΤΟ από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά είτε στρατηγική αντίδραση είτε πιο τοπική περιφερειακή αντίδραση. Και είναι ενδιαφέρον που οι δύο χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, η Νορβηγία και η Σουηδία για παράδειγμα, πρόσφατα έκαναν, ανέλαβαν κάποιες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις σχέσεις τους με το ΝΑΤΟ. Δεν θα ζητήσουν βέβαια ένταξη κανονική, γιατί γνωρίζουμε τις ευαισθησίες και τις πολιτικές πτυχές ε, μιας τέτοιας ενέργειας και των δύο χωρών, αλλά και οι δύο χώρες έχουν συνάψει συμφωνία εταιρική σχέσης με το ΝΑΤΟ στη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε πρόσφατα στην Ουαλία. Έτσι, με τις συμφωνίες αυτές μπορεί το ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει βάσεις στις χώρες αυτές, να κάνει γυμνάσια και να έχει κάποιες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό με τη διεύρυνση της συνεργασίας. Και αν θέλουμε πραγματικά να διαδραματίσουμε χρήσιμο και αποτελεσματικό ρόλο στην περιοχή, δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο σε διπλωματικές πτυχές, αλλά και σε θέματα ενεργειακής διαφοροποίησης. Γιατί μια άλλη αδυναμία των χωρών της περιοχής είναι ο βαθμός εξάρτησης ενεργειακής που έχουν από τη Ρωσία. Σε τελική πάντως ανάλυση ερχόμαστε στο θέμα της πολιτικής βούλησης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πόσο σοβαρά θα αντιμετωπίσουν οι χώρες μας το θέμα της ασφάλειάς τους. Γιατί μερικές χώρες περιόρισαν τις αμυντικές τους δαπάνες ε, και τις δυνατότητες ε, και τις ικανότητες ετοιμότητας και εγρήγορης που έχουν σε αντίθεση με τη Ρωσία που αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες και την ετοιμότητά της. Θα πρέπει η Βαλτική να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες γιατί οι σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ και οι νέοι μας σύμμαχοι ε, κάνουν νέες προσπάθειες. Υπάρχουν κάποια ελπιδοφόρα σημάδια ότι αυτές οι χώρες της Βαλτικής ε, τουλάχιστον θα λάβουν πιο σοβαρά υπόψη το θέμα της άμυνάς τους. Σας ευχαριστώ. Κύριος Νάρτ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω πάντως την έκπληξή μου, την κατάπληξή μου, γιατί εγώ θα περίμενα μια ανάλυση για τα βασικά σημεία που είναι σίγουρα το στρατηγικό, αλλά έχουμε και το κοινωνικό και τα κοινωνικά πτυχία, ε, τις κοινωνικές πτυχές και τις οικονομικές πτυχές. Τώρα μας παρουσιάσετε κάποιες ιαχές του πολέμου και παρουσιάσετε τη Ρωσία σαν να είναι ένα συνδυασμό Χίτλερ και Ατήλα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Σίγουρα δεν είναι όλες οι χώρες ίσες και υπάρχουν κάποιες προτιμήσεις, αλλά μερικές χώρες είναι πιο ίσες από άλλες. Κανένας δεν εκπλήσεται για τα στρατηγικά συμφέροντα που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο πολύ κυρίαρχο κράτος του Παναμά. Κανείς δεν διαρρήγνει τα ημάτια του. Και ε, ε, και σίγουρα κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος ε, ε, να παρήχε το κυρίαρχο κράτος του Παναμά τη διαχείριση της διόρυγας του Παναμά στη Ρωσία. Δεν νομίζω να θεωρούσε κανείς φυσιολογική μια τέτοια κατάσταση. Ενώ οι ΗΠΑ δεχόμαστε να υπερασπίζει τα συμφέροντά της με κάθε τρόπο, όπως έκανε η Σοβιετική Ένωση στο παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε τα στρατηγικά συμφέροντα των υπερδυνάμεων. Δεν λέω να τα αποδεχθούμε και να υποταχθούμε σε αυτά, αλλά για να τα καταλάβουμε τουλάχιστον, να τα συνειδητοποιήσουμε. Γιατί αν αντιμετωπίζαμε τη Ρωσία όποιος οποιαδήποτε άλλη χώρα που δεν έχει μια στρατηγική σημασία, για παράδειγμα την πατρίδα μου, την Ισπανία, νομίζω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος ε, βρισκόμαστε σε σύγχυση και δημιουργούμε μία ε, ιστερία αντιπαράθεσης ε, και πολεμικής ρητορικής. Σίγουρα έχουμε κάποιες ε, ζώνες σύγκρουση, αλλά ακόμη και στην εποχή του Στάλιν, κάποιες κόκκινες γραμμές δεν υπερκεράστηκαν, ακόμη και στην πολύ σοβαρή κρίση του Βερολίνου, ούτε με το Χρούστσεφ, με την εισβολή στη Τσεχοσλοβακία, με την ε, παρουσία στην Πολωνία. Ουδέποτε δεν ε, ξεπεράστηκαν συγκεκριμένε γραμμές και η αντιπαράθεση γινόταν στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, ποτέ όμως στην, ε, μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Μας παρουσιάζεται ένα σενάριο εισβολής, ε, επίθεσης, ε, επιδρομής στις χώρες του ΝΑΤΟ. Μα κάτι τέτοιο θα σήμαινε πυρηνικός πόλεμος. Και κατά τη γνώμη μου μια τέτοια πιθανότητα είναι τελείως παράλογη. Άλλο να έχει δραστηριότητες η Ρωσία σε κάποιες μαλαϊκές περιοχές, Ουκρανία, Γεωργία, πείτε τις όπως θέλετε, αλλά όχι στο ΝΑΤΟ. Αυτά τα, αυτές οι αρχές του πολέμου που ακούμε δεν νομίζω ότι έχουν θέση εδώ. Έχουμε υπογράψει στρατηγικές, ε, η Κίνα και η Ρωσία έχουν υπογράψει στρατιωτικές ε, στρατηγικές συμφωνίες. Μπορεί να δημιουργηθεί ένας ρωσοκινέζικος άξονας. Πώς βλέπετε μια τέτοια προοπτική. Επίσης, ποια είναι η επιχειρησιακή δυνατότητα ε, η, για, τη θύλακα του Καλίνικρατ, σε ό,τι αφορά το πολεμικό ναυτικό. Γιατί μόνο μία διέξοδο έχει στην Βαλτική η Ρωσία, το Κνόστατ. Ε, και έχει και μία έξοδο στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Μόνο μέσω του Βαλαδιβοστόκ έχει διέξοδο στην Ανοιχτή Θάλασσα και το Μούρμαρς. Ίσως στον Αρχάγγελο. Αλλά ελάχιστε είναι οι διέξοδοι της. Και τώρα εσείς μας μιλάτε για έλεγχο των στενών της Δανίας. Πραγματικά, μπορεί ως πολεμικό παιχνίδι να είναι ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, αλλά ως πραγματικό και ρεαλιστικό στρατηγικό σενάριο, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιανόητο και μιλήσατε για κάποια τροτά σημεία για την προπαγάνδα της Ρωσίας στις χώρες της Βαλτικής. Δίκιο έχετε. Σας ερωτώ όμως, για να δημιουργηθεί μια κατάσταση σταθερότητας θα πρέπει να έχουμε πρώτα κοινωνική σταθερότητα. Πιστεύετε ότι η διάκριση που υπάρχει ε, στις τοπικές κοινότητες, στις ρωσόφωνες τοπικές κοινότητες, στις χώρες της Βαλτικής και που συνεχίζεται αυτή η διακριτική μεταχείριση. Θεωρείτε ότι με μια τέτοια κατάσταση θα, θα δημιουργήσετε μια συνοχή στις χώρες της Βαλτικής και σε μια κοινωνική σταθερότητα που είναι το καλύτερο όπλο απέναντι σε οποιαδήποτε ρωσική προπαγάνδα. Μια κοινωνική συνοχή και σταθερότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρεκ Γιούρεκ. Α, συγγνώμη, πρώτα ο κύριος Σαφχάουζεν και μετά ο Μάρεκ Γιούρεκ. Παραχωρεί την σειρά του κύριο Σαφχάουζεν. Ευχαριστώ, Ζαν Λουκ. παραχώρησε τη σειρά του. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μια δια... εναλλαγή των διαφόρων απόψεων για να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εμπειρογνώμονες για τους πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους και να ευχαριστήσω και την πρόεδρο που ε, συμπεριέλαβε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πάνω από το 1 τέταρτο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κοντά στη Βαλτική και νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι στοιχειώδες θέμα αλληλεγγύης, γιατί αν δεν ενδιαφερθούμε για τη ζώνη αυτή και τις απειλές που αντιμετωπίζει, μια τόσο σημαντική ζώνη όπως είναι η Βαλτική, αν δεν δείξουμε τέτοιο ενδιαφέρον για τις ζώνες και τις περιοχές της Ένωσης, ε, πώς θα θέλουμε να λέμε την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, πραγματική Ένωση, αν αδιαφορούμε για την ασφάλεια των επιμέρους ζωνών της. Ο κύριος Χαβιέρ Νάρτ είπε ότι τέτοια υποθετικά σενάρια και τέτοιες απειλές είναι σημεία που ε, δεν είναι σχετικά και λογικά. Θα πρέπει όμως αντίθετα να σκεφτούμε σήμερα και να διαρωτηθούμε τι θα γίνει αν αντιμετωπίσουμε όντως τέτοια προβλήματα. Και ε, είδαμε τι προβλήματα είχαμε την τελευταία δεκαετία και στη Μαύρη Θάλασσα. Και μιλώ για την τελευταία δεκαετία, γιατί φαίνεται ότι μερικοί έχουν πολύ επιλεκτική μνήμη και ξεχνούν την προσάρτηση της Κρυμαία, αλλά πριν από 10 χρόνια, από λίγα από λίγα χρόνια, συγγνώμη, είχαμε και τον πόλεμο στη Γεωργία. Το ξεχνάτε αυτό. Δεν έχουμε μόνο το Don Έχουμε και ιστορικές εξελίξεις που προηγήθηκαν. Είπε ο κύριος Συνάρτη ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία με ίσο τρόπο όπως και τα άλλα κράτη. Έχουμε όμως ε, σημαντικό εταίρο τη Ρωσία και δεν θα πρέπει να διαφοροποιούμε τη την ρητορική μας ε, απέναντι στη Ρωσία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ρωσικές αρχές όπως οι ρωσικές αρχές αντιμετωπίζουν ε, τις ουκρανικές αρχές μήπως ή θα πρέπει να μιλήσουμε με την ίδια ρητορική που είχαν οι ρωσικές αρχές μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη γλώσσα που γνωρίζουν οι Ρώσοι, η ρωσική κοινή γνώμη και οι ρωσικές αρχές. Γιατί η Ρωσία κατηγόρησε τη Γεωργία ενώ ε, είχε κατεχόμενα εδάφη στη χώρα αυτή για πολλά χρόνια. Και μάλιστα σήμερα η Ρωσία χρησιμοποιεί μια φρασεολογία απέναντι στις ε, Ουκρανικές αρχές που ούτε καν τολμώ να την επαναλάβω. Η η Ρωσία δεν μπορεί να είναι κανονικός εταίρος ε, στη δημόσια, στην ε, διεθνή συνεργασία γιατί η Ρωσία ενεργεί με τέτοιο τρόπο που αρνείται οποιοδήποτε ρεαλισμό. Είμαι από μια χώρα που ε, ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση της σταθερότητας και της ειρήνης, ειδικά μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου και είναι και θέμα που αφορά μέσα και την κατάσταση μετά την ανάκτηση της ανεξαρτησίας μας. Γι' αυτό και είναι σημαντικό μαζί με τη Βαλτική να λάβουμε υπόψη και το θέμα της μαύρης θάλασσας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιο είναι ο βαθμός στρατικοποίησης και ποιες είναι οι απειλές από το θύλακα του Καλινιγκράτ. γιατί δεν χρησιμοποιούμε το Καλίνιγκραντ. Ε, συνήθως χρησιμοποιούμε ε, το Καλίνιγκραντ ε, και οι συνειρμοί που έχουμε με το Καλίνιγκραντ είναι δυστυχώς πολύ αρνητικοί με σφαγές και τα λοιπά. Δεν θα πρέπει πάντως εμείς μεταξύ μας να χρησιμοποιούμε τέτοιους ορισμούς, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Και νομίζω ότι συμφέρον είναι η αποστρατικοποίηση αυτής της περιοχής και νομίζω ότι θα πρέπει να, πούμε, να το δηλώσουμε αυτό με σαφήνεια, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κατάστασης που δημιουργήθηκε μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας. Μόνο η αποστρατικοποίηση του Καλίνιγκρατ θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Αλλιώ θα έχουμε συνεχή κατάσταση απειλής προς τις βαλτικέ χώρες και προς την Πολωνία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα να ζητήσω από τους εμπειρογνώμονές μας να συμπληρώσουν την ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας έδωσαν για τη Βαλτική και για την οικονομική ανάπτυξη της Βαλτικής, την οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας και πώς χρησιμοποιεί η Ρωσία σχέδια, σχέδια όπως το Nord Stream ως στοιχείο πολιτικής ε, αποσύνθεσης της συμμαχίας του ΝΑΤΟ αλλά και της ε, αποσύνθεσης και της ε, υπονόμευσης της Ευρωπαϊκής Ελληνικής. Ποια είναι τα τεχνικά στοιχεία της δημιουργίας του φυσικού αγωγού Nord Stream που μπορούν να τα εκμεταλλευτεί η Ρωσία για να οξύνει την αντιπαράθεση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσπαθήσει να μας διαιρέσει. Ιδιαίτερα να απομακρύνει ή να απομονώσει την Πολωνία και τις βαλτικές χώρες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και πιστεύω θα πρέπει, ότι σε όλα αυτά θα πρέπει να αντιδράσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πήγμη. Είναι σημαντικό να δείξει αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρωταρχικό στοιχείο της αλληλεγγύης είναι η αλληλεγγύη προς τις χώρες της Βαλτικής και η στήριξή τους στις προσπάθειες που κάνουν για να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία τους. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι ούτε στη Λετωνία ούτε στην Εσθονία δεν έχουμε διακριτική μεταχείριση των ρωσόφωνων κοινοτήτων. Οι απόγονοι ρωσόφωνων που έχουν παραμείνει στην Εστονία και την Λετωνία δεν πρέπει να πληρούν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στη, στον ενεργό πολιτικό βίο. Το πρόβλημα που απέμεινε είναι κάποιοι πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν στις χώρες αυτές από την ε, ρωσική, από τη σοβιετική ε, απεικιοκρατική εποχή. Δεν μπορείτε λοιπόν να, να κάνετε τέτοιους, ε, τέτοιες δηλώσεις για τέτοια διακριτική μεταχείριση και μόνο για να προκαλέσετε εντυπώσεις. Σίγουρα θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση στις χώρες της Βαλτικής και να τις στηρίξουμε και να μην επικαλούμαστε τέτοια επιχειρήματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, επιχειρήματα που ουσιαστικά χρησιμοποίησε με προκλητικό τρόπο στο Συμβούλιο της Ευρώπης η Ρωσία. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Βέβαια δεν έχουμε και πάρα πολλού εδώ συναδέλφου, το οποίο είναι απογοητευτικό για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. για θέμα άμυνας και ασφάλεια. Αλλά αναρωτιέμαι όσον αφορά το τι επιζητούμε. Με την πτώση του τείχους άρχισα να αφοσιώνομαι στο τι γίνεται ως προς τον, τον πολυσεβικισμό, πώς μπορούμε δηλαδή να έχουμε κάποιο είδους άμυνα ευρωπαϊκή, γιατί πάρα πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει αληθής βούληση ούτω ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή άμυνα. και στη χώρα μου τη Γαλλία έχω ασχοληθεί με τα θέματα άμυνας και ασφάλειας αλλά μιλώ γενικότερα για την Ευρώπη η Γαλλία που είναι μια πυρηνική ανεξάρτητη δύναμη και από την άλλη μεριά η Ρωσία. Έχουμε λοιπόν στην Ευρώπη δύο τέτοιες ε, ανεξάρτητες αυτόνομες ε, δυνάμεις. Επομένως, με το που έπεσε το τείχος, το ΝΑΤΟ πήρε την θέση που ε, άφησε η ανικανότητα η Ευρωπαϊκή να οικοδομήσει μια τέτοια άμυνα. Οπότε και αυτό πάσχησα να κάνω, δούμε πώς θα έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη σε αυτό, γιατί θεωρήσαμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν θεμητά συμφέροντα. Αλλά όμως και η Ευρώπη έχει θεμητά συμφέροντα. Και τα αμερικανικά συμφέροντα πολλέ φορέ ταυτίζονται με τα δικά μας, αλλά όχι αναγκαστικά. Γιατί έχουμε δικά μα ευρωπαϊκά θέματα. τα αμερικανικά συμφέροντα είναι να κοπεί η Ευρώπη στα δύο. Το έχει γράψει ο Μπρεζίνσκι. Έχουν τον τρόπο. Και καταλαβαίνω, γιατί πίσω από το δόγμα του Ατλαντισμού υπάρχει μια ισχύς που μπορεί να αντισταθμίσει, να αντιμετωπίσει την Κίνα. Οπότε πρέπει να κοπεί η Ευρώπη από τη Ρωσία για να μην υπάρχει τέτοιου είδους άξον ευρωπαϊκός, υπηρετικός που αφορά τα ενεργειακά. Το 1995 είχα μιλήσει με τον πρόεδρο Κούσμα και μου εξηγήθηκε τι κάνανε οι Αμερικανοί τότε. Είναι παλαιό το σχέδιο, οπότε ναι, όντως οι Αμερικάνοι πάνε να βρουν Λιθουανούς, Πολωνούς, ε, που, γιατί υπάρχει πολωνική διασπορά μεγάλη στην ε, Αμερική ε, οι Αμερική, οι ονειρεύονται την ε, κάποτε μεγάλη Πολωνία και βρίσκουν ε, συμμάχους οι Αμερικανοί όμως τι γίνεται, πού, πού θα μας οδηγήσει αυτή η συνεχής πολιτική της επιθετικότητας γιατί έχετε εφετηρία το ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος. Αλλά για μπείτε στη θέση των Ρώσων που εκείνοι θεωρούν ότι το ΝΑΤΟ είναι ο επιτιθέμενος. Ο Γκορμπατσόφ το είπε όταν έπεσε το τείχος. Δεν θέλουμε επέκταση του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτή την Ενωμένη Ευρώπη τη χρωστούμε στον Γκορμπατσόφ. Τη διευρυμένη Ευρώπη. Και ενώ δεν συμφωνεί, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, τον υποστηρίζει τον Πούτιν. Τι λέει ο κύριο Σόρο, Λέει να ενωθεί η Ευρώπη και να κάνει έναν ε, πόλεμο κατά της Ρωσίας. Μα πού θα μας οδηγήσουν όλα αυτά. Να σας πω. κάποια στιγμή θα αντιδράσει η Ρωσία. Ή θα πρέπει να μπούμε σε μια πυρηνική σύγκρουση, οπότε πιστέψτε με θα είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε μόνο να χάσουμε έχουμε ως Ευρώπη. Και τι θα απομείνει Ασία, Κίνα, θα, θα υπάρχουν αρκετοί και έτσι θα φτιαχτεί ένας καινούριος κόσμος. Αλλά η Δύση, η Δύση από αυτόν τον ολοκληρωτικό πόλεμο μόνο χαμένη θα βγει. Θα σας το λέω φίλοι Πολωνοί, φίλοι από τις βαλτικές χώρες σας το λέω φιλικά. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει με αυτά τα μικρά παιχνίδια επιθετικότητας. Είμαι Γάλλος. και όταν ε, την επαύριο ανέβουμε στην εξουσία θέλουμε να βγούμε από τον ΝΑΤΟ όπως το θέλαμε ανέκαθεν στη Γαλλία. Τίποτα δεν θα γίνει. Οπότε η λύση ποια είναι γενικός, γενικευμένος πόλεμος ή αυτή η κατάσταση της επιθετικότητας που δεν μας οδηγεί πουθενά είναι ένα αδίέξοδο και το γνωρίζετε. Γιατί έτσι όπως πάτε γυρεύοντας, επιζητείτε πόλεμο, θα τον βρείτε μπροστά σας τον πόλεμο. Ja chciałem odpowiedzieć na to, mm, na wypowiedź pana Schaffhausena. Ναι, εγώ θα ήθελα τώρα... Θα ήθελα λίγο να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος. Κοιτάξτε, δεν σας αντιλαμβάνομαι πλήρως. Η Ευρώπη εγγυάται υποτίθεται και την ασφάλεια της Γαλλίας και άλλων χωρών. Αλλά μην ξεχνάμε την ασφάλεια της Λετωνίας, της Λιθουανίας, χωρών της Βαλτικής. Η Βαλτική είναι μια ευρωπαϊκή θάλασσα. Εσείς το παρουσιάζετε σαν να υπάρχει σύγκρουση ή παρουσίας. Όχι, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Το θέμα είναι η ασφάλεια των χωρών της Βαλτικής. Ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτά τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Και όταν μιλούμε για ε, επίθεση, ας μην ξεχνούμε και την ιστορία. Ε, και ας μην κάνουμε με τα στραβά μάτια. Ξέρουμε ποιος στην περιοχή αυτή έχει επιθετικές στάσεις. Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα, τη Ρωσία, που είναι ε, η διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης, ε, μιας ε, ένωσης που κρατούσε στη, στη δουλεία υπό το ζυγό της στη μισή Ευρώπη. Και βέβαια ακούσαμε μετά τη διάλυση ότι το μεγαλύτερη ε, για πολιτική τραγωδία ήταν η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι τέτοιοι ισχυρισμοί είναι δεικτικοί της τάσης και γνωρίζουμε τον ιστορικό ρόλο της Γαλλίας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και εσείς ως Γάλλος γνωρίζετε κάλλιστα ε, το ρόλο της Γαλλίας και ανεξάρτητα από αυτό γνωρίζουμε ότι και στο μέλλον θα έχει γεωστρατηγικό ρόλο η Γαλλία και ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη. Και να μην ξεχνά και τους ιστορικούς δεσμούς που έχει η Γαλλία με πολλές από τις χώρες της περιοχής και γι' αυτό να λάβει υπόψη την ασφάλεια και την ευημερία και τη μελλοντική ανάπτυξη αυτών των χωρών. Απευθύνω λοιπόν έκκληση, δηλαδή υπόψη και ο συνάδελφος ή πρόεδρος. Θα ήθελα κι εγώ ως μέλος της Υποεπιτροπής να λάβω το λόγο για να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις, ε, χωρίς ε, να μακρηγορήσω όμως, για να μην στερήσω από τους καλεσμένους μας ε, τη δυνατότητα και το χρόνο για να απαντήσει. Σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έγιναν για το θέμα, νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ επίκαιρο και εντάσσεται κάλλιστα στις ε, αρμοδιότητες της υποεπιτροπής μας, γιατί είμαστε υποεπιτροπή ασφάλειας και άμυνας. Και το θέμα της πειρατείας στο κέρας της Αφρικής εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας και, και η ασφάλεια της Βαλτικής είναι ακόμη πιο σημαντικό θέμα, γιατί η Βαλτική είναι εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πολύ περισσότερο είμαστε αρμόδιοι για το θέμα αυτό. Και Έχουμε πολλές χώρες μέλη που βρίσκονται στην περιοχή αυτή που ανέκτησαν το 1989 την ανεξαρτησία τους και με την υποστήριξη του Πάπα Ιωάννη Παύλου του δεύτερου κύριε Σαφχάουζεν. Αυτό είναι αλήθεια και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη μεγάλη υποστήριξη που μας παρήχε τότε ο Ιωάννης, Πάπας, Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος και δεν είμαστε ε, υγειονομική, υγειονομικός κλειός. Είμαστε ανεξάρτητες χώρες και φυσικά δεν θέλουμε να γίνονται πράγματα πάνω από το κεφάλι μας και να υφιστάμεθα απειλές. Και πιστεύω ότι ακριβώς η υποεπιτροπή μας είναι το κατάλληλο φόρουμ για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα των απειλών και της κοινή αντιμετώπισης τους από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου και αν λαμβάνουν χώρα αυτές οι απειλές και η εσωτερική αλληλεγγύη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερτερεί κατά τη γνώμη θα έπρεπε να υπερτερεί της οικονομικής αλληλεγγύης εφόσον έχουμε απειλή της ασφάλειας και εδώ έχουμε πολλά σχέδια συμφωνίες και εταιρική σχέσεις ε, με τη Ρωσία που ακριβώς ε, επηρεάζουν ε, άμεσα την ασφάλεια των χωρών. Γι' αυτό και έκρινα σκόπιμο και κατάλληλο να συμπεριλάβω αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είμαστε ανεξάρτητες χώρες, οι χώρες της Βαλτικής και έχουμε τεράστια, πολύ πλούσια πείρα ε, συμβίωσης ε, πολύ κοντά σε μία υπερδύναμη όπως είναι η Ρωσική Ομοσπονδία και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εμείς επιθετικοί επιθετικότητα ήταν η στάση που έδειξε η Ρωσία όταν εισέβαλε στην ε, κυρίαρχη Γεωργία και ακόμη περισσότερο όταν προσήρτησε την Κρυμαία. Και νομίζω ότι ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους ήταν πολύ σκόπιμο να συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας γιατί έχουμε και άλλα σημεία μετά να συζητήσουμε. Πάρα πολύ ζωντανή συζήτηση, Πρόεδρε. Και αυτό μας δείχνει ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Πέραν του αν κάποιοι βουλευτές είναι υπέρ, κάποιοι κατά. εγώ ο κύριος Τομάς τη λέμε ε, σε σχέση με αυτά. Κάποια από αυτά που σαν αποτελούν μάλλον ε, δηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα και δεν είναι τόσο ε, συγκεκριμένα. Ορισμένοι αναφέρθηκαν στο Καλινιγκράτ που οπωσδήποτε είναι ζήτημα σημαντικό. ήδη τώρα έχει περισσότερο ρωσικό στρατό παρά όσο στρατό έχουν όλες οι βαλτικές χώρες μαζί. Να, επομένως, πώς έχουμε την στρατηγική ισορροπία εκεί και το σούτο μάλλον κατά πόσο καθώς το, χρησιμοποιείται το καλύνδρατα από πλευρά Ρώσων ως ε, μοχλός πίεσης. Κάντε κάτι, αλλιώς θα κάνουμε εμείς εκείνο, λένε οι Ρώσοι. Στο λιμάνι, με τους πυράβλους, ε, θα, θα, σας κλείσουμε τη, την πρόσβαση στη θάλασσα κλπ. Γι' αυτό και προβληματίζουν πολύ οι εκεί εξελίξεις και τις παρακολουθούμε από κοντά. Σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο κύριος Φανόρντιν, δηλαδή, σε ποιο βαθμό τα κράτη εκεί παίρνουν στα σοβαρά το θέμα της ασφάλειας, τα είπαμε. Είπαμε ότι αυξάνουμε τις αμυντικές δαπάνες. Και βέβαια η οικονομική κρίση 2009 και 2010 μας έπληξε στην Λετωνία, οπότε και τότε είχαμε συρρήγνωση των αμυντικών δαπάνων. Πάντως, ε, τώρα η κυβέρνηση και το κοινοβουλίο μας ε, επιμένουν στο μέτωπο αυτό και αυτή η αύξηση θα αντικατοπτρίζεται στον επόμενο προϋπολογισμό του χρόνου. Κάτι που ρωτήθηκε από τον κύριο Νότ για την Ρωσία. Το αντίθετο ισχύει κύριε. Εμείς τα κράτη της Βαλτικής, είμαστε μέλη της ε, Ατλαντικής Συμμαχίας και της Δύσης, θεωρούμε ότι η Ρωσία είναι ένα έθνος ίσο με μας. Και η απομάκρυνση μας από, από κάποιες συνθήκες όπως σας ανέφερα αυτό έφερε κάποια απομάκρυνση, επομένως κάποια αποξένωση και είπαμε όμως ότι από την άλλη μεριά έχουμε τον ακρογωνίο λίθο της ε, ευρωπαϊκής ασφάλειας. Δεν, το, δεν αποξενωθήκαμε όμως εμείς από αυτή την αρχιτεκτονική της ασφάλειας. Η Ρωσία το έκανε και θυμάμαι πριν από καιρό, τη δεκαετία του 70, διάφορα κράτη στο βόρειο ημισφαίριο συμφώνησαν στο Ελσίνκι να μην παραβιάζουν την καθιστική ατάξη, ας πούμε, πέραν των υγειοστρατηγικών μεταβολών. Είδατε τι έγινε με την κατάληψη της Κρυμαίας. Είδατε τι έγινε στην Αμπχαζία, τι έγινε στην Νότια Ρωσετία, τι έγινε με τα κράτη αυτά τα οποία απεσχίστησαν. Και θα το βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα κάποιος κάνει τόσο σημαντική παραβίαση. Γινόμαστε μάρτυρες της παραβίασης ενός ε, μιας αρχής από τις πιο βασικές, τις πιο σημαντικές στη μεταπολεμική εποχή. Αυτό είναι η ενσυχία για το μέλλον. Είναι κατακλείδη να σας πω ότι συμφωνώ για το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ελληνικής. Και όπως προείπα, οι χώρες της Βαλτικής έχουμε επιδείξει αλληλεγγύη προς άλλες περιοχές της Ευρώπης έχουμε ανταποκριθεί στις ανάγκες των συμμάχων μας. Επιχειρήσει στο Αφγανιστάν, η καταπολέμηση της πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό, η υποστήριξή μας για μια σειρά προβλημάτων είτε στο Μαλί είτε στην Κεντρική Αφρική Πάντοτε ανταποκρινόμαστε όποτε μας καλούν κάποιοι. Αλλά τώρα ήρθε να καλέσουμε εμείς σε βοήθεια. Και αυτό πια δεν είναι ένα αστείο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για το Καλίνιγκραντ που αναφέρθηκε κάνα δύο φορές. Αυτή τη στιγμή στο Καλίνιγκραντ υπάρχουν τρεις ταξιαρχίες, ε, τρεις μηχανοκίνητες ταξιαρχίες και ε, εξοπλισμός για δύο ακόμα μεραρχίες ε, όταν έρθει το προσωπικό. Και μάλιστα το 2006 Ρώσοι και Λευκορώσοι εκπαιδεύονταν για την επάνδρωση περαιτέρω μονάδων. Τώρα το ερώτημα είναι αν το Καλίνιγκραντ θα μπορέσει να αποτελέσει προκεφύρωμα εισβολής ή απλά θα είναι ένα αγκάθιστα μετόπιστεν ε, που θα κυρώνει τη δυνατότητα ελέγχου της Βαλτικής σε περίπτωση εκτοπραξιών του. Άλλα σημαντικά στοιχεία. Η αεράμινα του Καλίνιγκραντ μπορεί να ακυρώσει τον αεροπορικό έλεγχο της Νότιας Βαλτικής. Δεύτερον, κάποιες φορές είδαμε δραστηριότητα ε, που ήταν η ανάπτυξη βλημάτων Ισκάντερ στο Καλίνιγκραντ. Το εάν είναι εκεί τώρα ή όχι δεν έχει τόση σημασία γιατί τα βλήματα μπορούν να μεταφερθούν εκεί σε 24 ώρες. Και όπως ξέρετε οι περισσότεροι κεντρική και ανατολική Ευρώπη είναι εντός του σε αυτών των βλημάτων. Είναι ευλήματα, επαναλαμβάνω, που μπορούν να φέρουν ε, τακτικές πυρηνικές κεφαλές. Αυτά περί Καλίνιγκραντ. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κ. Ζέμκε για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου θα πρέπει εδώ να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της αποφασιστικότητας, της πυγμής και της αποφυγής της κλιμάκωσης. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς βλέπει ο, η άλλη πλευρά το θέμα. Και μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι η Ρωσία ε, εξετάζει όλα αυτά υπό τη σκοπιά του ψυχρού πολέμου. Οπότε θα πρέπει να δείξουμε πυγμή, αποφασιστικότητα και να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να αντιπαραταθούμε σε μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Βέβαια, μια τέτοια πυγμή και αποφασιστικότητα ίσως οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί σε περίπτωση παραβίασης αέριο χώρου θα πρέπει να στείλουμε ε, αεροπλάνα που θα αναχαιτήσουν τους παρήσακτους ε, θα πρέπει να δούμε ε, τι κάνει, τι σκοπό έχει η πλευρά που προκαλεί αυτή την κλιμάτωση και που είναι υπεύθυνη για την ε, διατάραξη της ασφάλειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές πτυχές ή τις ε, πτυχές ασφάλειας που σχετίζονται με την κατασκευή του Nord Stream. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που έκανε ένα σουηδικό think tank για την κατασκευή αυτού του αγωγού φυσικού αερίου και που λέει ότι ίσως έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια. Ε, επίσης κάποιες ε, δραστηριότητες ε, κατασκοπικές ή συγκέντρωσης ε, πληροφοριών. Ή να χρησιμοποιηθεί η κατασκευή του Nord Stream ως πρόσημα για την ενίσχυση της στρατιωτικής κινητικότητας. Σας μίλησα προηγουμένως για τον υβριδικό πόλεμο. Τι τις υβριδικές ενέργειες. Επίσης, για αυτά που είπαν ο κύριος Νάρτ και ο κύριος Σαφχόιζεν. μίλησαν για διπλά μέτρα και σταθμά. Γιατί είπαμε σε προηγούμενο πόλεμο ήμασταν πιο επίκης γιατί δεν ε, ξεπέρασε η άλλη πλευρά κάποιες ε, σημαντικές κόκκινες γραμμές. Αλλά νομίζω απάντησε εύστοχα στα σχόλια αυτά η πρόεδρος Φωτίγκα. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους δύο εμπειρογνώμονές μας ε, για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις και σας ευχαριστώ θερμά που παραμείνατε και παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση και χωρίς διάλειμμα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους επόμενους μας καλεσμένους. Έχουμε καταρχήν την κυρία Πάολα Ιμπεριάλε, εκπρόσωπο της Ιταλικής Προεδρίας είναι συντονίστρια στο, στο Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα ναυτιλίας και θα μας παρουσιάσει το σχέδιο δράσης για την στρατηγική ασφάλεια της ναυσιπλοείας που αποτελεί προτεραιότητα και μάλλον πρωτοβουλία της Ιταλικής Προεδρίας. Ο δεύτερος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ρούντολφ Ρόι, που είναι τμήματάρχης ε, στην αρμόδια διεύθυνση της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και είναι αρμόδιος για θέματα ασφάλειας, πολιτικής ασφάλειας, όχι ασφάλειας και κυρώσεων που είπα εσφαλμένα προηγουμένως και τρίτη καλεσμένη, κυρία Μπεάτε Γκμίντερ, που είναι τμήματάρχης ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής με ειδικότητα στην Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Ιμπεριάλε Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι, κυρία Ιμπεριάλα, και αν έχετε χρόνο να παραμείνετε και για να ακούσετε τις ερωτήσεις και να δώσετε απαντήσεις, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ πιεσμένο χρονοδιάγραμμα. Θα δούμε πόσο μπορείτε να παραμείνετε στη συνεδρίαση. Πρώτα λοιπόν η κυρία Πάολα Ιμπεριάλε από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά ο κύριος Σερό και μετά η κυρία Κμίντερ. Ε, Καλημέρα σας. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Πρόεδρο, διότι μου δίνει την ευκαιρία να σας ανακοινώσουμε το έργο της ε, Ιταλικής Προεδρίας αλλά και της Ελληνικής που προηγήθηκε. Τι έγινε με την ασφαλεία της θάλασσες Και ειδικότερα στην Μεσόγειο έχουμε εξασφαλίσει μια συνέχεια στην πολιτική και ακόμα δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που χάνονται στις θάλασσες και έχουμε ξαναεπισκεφτεί την υποεπιτροπή σας και αναφερθήκαμε στο έργο μας αλλά και στην μελέτη εκείνη την οποία είχε αναλάβει η Επιτροπή σας για τις γεωστατηγικές εξελίξεις στη θάλασσα. Ήταν ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή των απόψεων για τις επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, διαπιστώθηκε η ανάγκη του να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική. Είχαμε επίσης και την έκθεση Γκόμες που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Επίσης θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για αυτό το υλικό αλλά και για την ε, αγαστή συνεργασία διότι ανεξαρτήτως του ότι έληξε μια θητεία, ξεκίνησε μια καινούργια για το κοινοβούλιο, η συνεργασία μας είναι καλή και έτσι μπορούμε να έχουμε μια πολιτική ούτως ή πριν καθοδήγηση αυτά τα οποία κάνουμε. Οπότε και έτσι καλύπτουμε τις ε, προσδοκίες, τις προοπτικές μας για το μέλλον. Θα πρέπει βεβαίω να ευχαριστήσουμε και την Ελληνική Προεδρία, γιατί και εκεί μπήκε ένα λιθαράκι στο έργο μας αυτό για την ε, ασφάλεια αλλά και την ε, άμυνα για τη θάλασσα. Επίση, πάρα πολύ χρήσιμο ε, ήταν εκείνε οι δηλώσεις, οι κοινέ τι οποίε κάναμε μετά τη συζήτησή μα και ήταν πολύ καλή συνεργασία των άλλων προεδριών με την δική μας. Επίσης έτσι μπορέσαμε να έχουμε κάποιες ε, κοινέ συναντήσεις ε, ε, για τη χάραξη της πολιτικής και έτσι μπορούσαμε να φτάσουμε σε κάποια αποτελέσματα οπότε όλοι οι πρωταγωνιστές είναι στη χάραξη αυτή της πολιτικής. Αυτή η κοινή διαδικασία, η κοινή συνεργασία, η κοινή εργασία μας έδειξε το τι θα πρέπει να γίνεται σε σχέση με το χάρτη πορεία που αποφάσισαν οι επικεφαλεί κρατών για κυβερνήσεων το Σεπτέμβριο Νομίζω ότι γνωρίζετε περί την πρόκειται. Πάντως, τον Ιούνιο εγκρίθηκε η πολυκλαδική στρατηγική μας και διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ πολιτικών και σταθιωτικών υπηρεσιών για τη θάλασσα. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι κατά θάλασσα, το εργονομένο έγκλημα, οι φραγμοί στην ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αλλά επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις απειλές κατά του περιβάλλοντος. Χρειάζεται και μια διακυβέρνηση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το διεθνές δίκαιο. Και θα πρέπει να εμπλακούν και οι εθνικές αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την ασφάλεια στη θάλασσα. Κάτι το οποίο το λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε όταν ε, εκπονούμε ένα πρόγραμμα δράσης. Ε, θέλουμε να υπάρχουν και καινούργιες δομές αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ό,τι ήδη έχουμε στα χέρια μας σαν μέσα πολιτικές. Θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στην κοινούς στις πρωταγωνιστές στην παρουσία μας στη θάλασσα, να προβληθούμε περισσότερο και η Ιταλική Προεδρία από αρχές Ιουλίου ε, ανέλαβε να οργανώσει μια διάσκεψη. Αυτή η διάσκεψη έγινε σε μια στρατιωτική βάση, ναυτική στρατιωτική βάση και έτσι και όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρήσαμε ότι μπορούν να βοηθήσουν το Συμβούλιο στο έργο του. εν όψη και του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου, οπότε και θα υψηλογιστεί το έργο μας, θα ολοκληρωθεί με ένα έγγραφο εργασία. και έχουμε ήδη συντάξει το πέμπτο και ελπίζουμε τελικό σχέδιο κειμένου σχετικά με αυτό. Έχουμε 130 δράσεις που αφορούν το τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει από πλευρά κομισιών, κρατών μελών, Θα ήθελα τώρα να σας πω κάποιες σκέψεις μου σε σχέση με την εφαρμογή της πολιτικής και το να συμπορευτεί μαζί μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε να εξετάσουμε τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ, να έχουμε νέες δομές να δούμε τη σχέση μεταξύ ιστορικών και εξωτερικών ε, παραγόντων. Όλα αυτά τα λέμε στο έγγραφο που σας προανέφερα και αυτό το πρόγραμμα δράσης καλύπτει και τις, ε, την εμπλοκή των στρατιωτικών οπότε θέλουμε να έχουμε μία σφαιρική προσέγγιση και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπλακούν όλα ένα και περισσότεροι για να εφαρμόσουμε την πολιτική μας, να εντοπίσουμε τις σχετικές προκλήσεις, οπότε και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για εφαρμογή αυτού του προγράμματος δράσης. Να συνεργαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο σε σχέση με τις αρχές που προανέφερα. Να λαμβάνουμε βέβαια υπόψη τις δημοσιονομικές πιέσεις που έχουμε όλοι μας σε σχέση και με τις εθνικές προτεραιότητες. να δούμε τι ευκαιρίε πρέπει να εκμεταλλευτούν, όπω λέει το πρόγραμμα δράση, γιατί οποτεδήποτε είναι δυνατόν θα πρέπει να έχουμε ως βάση τα όσα θετικά ήδη έχουμε πετύχει. Θα πρέπει τις υπάρχουσες δυνατότητες να τις εκμεταλλευτούμε. Τα προγράμματα, το, το πρόγραμμα για την διαλειτουργικότητα και όλα τα άλλα προγράμματα τα οποία ήδη λειτουργούν τα χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, κέντρα εκπαίδευση, αριστείας, έρευνας, επίση και να μην έχουμε επικάλυψη ενεργειών. Έρευνα, κατάρτιση, εκπαίδευση. Έτσι θα εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν και να μην υποτιμήσουμε το, τη βιομηχανική πτυχή αυτού του προγράμματος δράσης. Η, η πολιτική μας, όλα και περισσότερο βέβαια γενικότερα στην Ένωση, έχει να κάνει με ανάπτυξη και απασχόληση και γι' αυτό να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα δράσης και γι' αυτό να μπορέσουμε να έχουμε μια εφαρμογή που να έχει καλή σχέση κόστους αποτελέσματος και θα πρέπει να μπορέσουμε να παράσχουμε την ασφάλεια που θέλουμε και να μην ξεχνούμε πόσο σημαντική είναι η εταιρική σχέση η ευρωπαϊκή, κάτι το οποίο αφορά και αυτό το πρόγραμμα δράσης. Και έτσι να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη και την προσαρμογή του πρόγραμματος δράσης στις μελλοντικές εξελίξεις. Και μόλις εγκριθεί αυτό το πρόγραμμα, αυτό θα είναι μια καινούργια αφετηρία, γιατί θα ξαναπευθούμε σε εσά όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος και να δούμε επίσης ε, σε ό,τι απορίες έχετε πώς θα σας δώσουμε τις απαντήσεις. Now, Mr. Roy, please. Ευχαριστώ, κύριος Ρόι. Sorry, uh, I was told at very short notice I have to, to, to change the order and now... Τελευταία στιγμή μου είπαν πρέπει να αλλάξουμε τη σειρά. Κλείνει το μικρόφωνο της Πρόεδρου τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να είμαι εδώ. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε πριν από έξι μήνες επί ελληνικής προεδρίας και χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε η κυρία για την ε, Ιταλική Προεδρία και τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ελπίζοντας λοιπόν να μην επαναλάβω τα όσα είπε η Πάολα, νομίζω πως σημασία έχει να αντλήσουμε αυτό το δίδαγμα. Η συνεργασία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ε, δρόντων ε, των μάλλον στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική μπορεί να είναι πάρα πολύ θετική, να έχουμε συνεργασίες, αποτελέσματα και βεβαίως πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο δράσης και υπάρχει τώρα το σχέδιο δράσης με πολλές δράσεις αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο και πολιτική ε, βούληση. Και βεβαίως ε, θα ήθελα και εσείς ε, να στηρίξετε το μήνυμα της συνεργασίας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών ε, μέσω της συζήτησης του σχεδίου αυτού δράσης σε άλλες επιτροπές. Καλό είναι να το αγκαλιάσετε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό. Ε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και για μας ε, και ε, στα κράτη-μέλη και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι ένα εγκάρσιο προϊόν που πρέπει να το εξηγήσουμε σε όλους τους εμπλεκομένους και απαιτείται και στήριξή τους. του λεχθέντος είναι σαφές πως δεν ε, έχουμε πανεφεύρει τον τροχό. Βασιζόμαστε σε αυτά που έχουμε ήδη επιτύχει. Είναι σημαντικό αυτό. Δίνουμε μια συμπληρωματική πίνελιά να προσθέσουμε και τη δική μας προοπτική αλλά η κάθε δράση έχει ένα κέντρο βαρύτητας ας πούμε αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει και να εφαρμοστούν αυτά στην πράξη. Να σας δώσω τρία-τέσσερα παραδείγματα από τις δέσμες της εργασίας μας. Το ένα είναι ε, η κοινοποίηση πληροφοριών, υπάρχει ένα σχετικό περιβάλλον που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη με βασική ιδέα να μοιραζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες των αρχών, των αρμοδιών αρχών λιμενικό, νοριοφύλακε, πολεμικό ναυτικό, επόπτες αλληλείας, τελωνιακούς, ε, όλοι αυτοί παράγουν δεδομένα, τα επεξεργάζονται και γνωρίζουν. Αν τα μοιραστούμε αυτά, γνωρίζουμε τι συμβαίνει στη θάλασσα και μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τις θάλασσές μας και θα προστατεύονται οι πολίτες μας. Πρέπει πάντα να το έχουμε κατά νου αυτό. Βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, αλλά το να υπάρχει μια στρατηγική πολιτική σκέπη, θα έλεγα, της ε, ευρωπαϊκής ε, θαλάσσιας στρατηγικής θα βοηθήσει στην εφαρμογή του. Τώρα, για την αξιολόγηση κινδύνου. Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι παρόμοιο όταν μιλάμε για την ανάλυση κινδύνου. Κάτι το οποίο κάνει κάθε δημόσια αρχή μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις αναλύσεις, να διευρύνουμε και πάλι την γνωσιολογική μας βάση. Εγώ θα έλεγα ναι. Και είναι κάτι βεβαίως το θετικό, αλλά πρέπει να ξεκινήσει. Ένας άλλος τομέας συνεργασίας που είναι πάρα πολύ σημαντικός είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση. Υπάρχει πράγματι διάθεση συνεργασίας, έχουμε ε, και διαφορετικούς εκπαιδευτικούς φορείς ε, για την σταδιοδρομία. Βεβαίως μιλάμε κυρίως για το δημόσιο όταν μιλάμε για την ασφάλεια των θαλασσών και έχουμε επίσης ένα δίκτυο λιμενικών. ή λιμενικών αρμοδιοτήτων ε, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει ας πούμε και τελωνιακούς, ε, συνοριοφύλακες ε, και τα λοιπά που ασκούν αρμοδιότητες λιμενικού σώματος. Να υπάρχει μια κοινή εκπαίδευση και κατάρτιση και πιθανώς κάποιο κοινό σύστημα ευρωπαϊκών προσόντων. Αυτές είναι κάποιες συγκεκριμένες ε, ιδέες. Βεβαίως ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ε, η Κομισιόν στήριζε το σχέδιο αυτό δράσης. Ευχαριστούμε και την mm. Προεδρία για την καλή συνεργασία. Ελπίζουμε να ενδιαφέρει και το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να το παρακολουθείτε και να το ενσωματώσετε και στο έργο άλλων επιτροπών και να το δουν και οι συναδελφοί σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Πολύ καλή παρουσίασή σας κύριε Κμίντερ. Ο κύριος Ρόι τώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω, γιατί είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η στήριξη της Επιτροπής σας και ο ηγετικός της ρόλος στο θέμα αυτό, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο εξάμεινο, όπως είπαν οι κυρίες Ιμπεριάλε και Γκμίντερ. Θέλουμε αυτή τη δέσμευση, αυτή τη στράτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και στο μέλλον. Γιατί ακόμη και με την έγκριση του σχεδίου δράσης που ευελπιστούμε ότι θα λάβει χώρα το Δεκέμβριο δεν θα έχουμε διαθετήσει τα πάντα. Πολλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν και μετά την υιοθέτηση του σχεδίου δράσης. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ήταν μια κοινή προσπάθεια των Προεδριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που όπως σας είπα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Και μάλιστα η φετινή χρονιά ήταν πολύ επιτυχή σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην αυσιπλοεία. Είχαμε και πρόσφατα, στις αρχές του έτους μάλλον, την ε, κοινή ανακοίνωση κατόπιν τη στρατηγική που εξήγηλε το καλοκαίρι η Ελληνική Προεδρία και τώρα περιμένουμε διακαώς και το σχέδιο δράσης αν κάνετε τη σύγκριση με την κατάσταση πριν από ένα χρόνο, θα δείτε ότι πραγματικά επιτελέσαμε εντυπωσιακή πρόοδο. Τώρα, για το σχέδιο δράσης καθ' αυτό. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι ένα έγγραφο όχι στατικό, μια πολιτική όχι στατική. Το έγγραφο είναι μία ζωντανή πρωτοβουλία, δεν είναι μόνο ένα έγγραφο. Θα πρέπει να εφαρμοστεί εμπράκτος και να τύχει και στενής παρακολούθηση στο μέλλον. Μάλιστα, για τα σχέδια δράσης έχουμε χρονοδιαγράμματα και για βραχυπρόθεσμες αλλά και, και για μέσο και μακροπρόθεσμες δράσεις. Όπως ε, ακούσαμε υπάρχουν πτυχές εξωτερικών σχέσεων, ε, ανταλλαγής πληροφοριών, ανάπτυξη των ικανοτήτων, διαχείριση κινδύνων, έρευνας και κατάρτισης. Είναι διαφορετικοί αυτοί οι τομείς, αλλά άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Για παράδειγμα, γίνουν γυμνάσια για την ε, ασφάλεια της ναυσιπλοείας Αυτά τα γυμνάσια φυσικά έχουν και μια εξωτερική πτυχή, αν συμμετέχουν σε αυτά και κάποιοι εξωτερικοί εταίροι μας, αλλά ε, είναι και θέμα που άπτεται της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η, η πιθανή χρήση διαστημικών ικανοτήτων, όπως τα προγράμματα Κοπέρνικος και Γαλιλαίο, Αυτά φυσικά συμβάλλουν στην ετοιμότητα, την εγρήγορση και την παρακολούθηση, αλλά είναι τμήμα και τη συζήτηση για τη διπλή χρήση, στρατιωτική και πολιτική. Και θεωρούμε ύψιστη προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου που θα συμπεριλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές, όπως είπαν οι προλαλήσεις σας. Θα επικεντρωθώ τώρα σε τρία βασικά σημεία θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν ξεκινούμε εκ του μηδενός, αλλά αξιοποιούμε το υπάρχουσες δράσεις. Η επιχείρηση Αταλάντη, για παράδειγμα, αναφέρθηκε ως παράδειγμα, αλλά και προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σημαντικές ε, θαλάσσιες ε, λεωφόρους για τη δημιουργία ικανότητων. Και ο συντονισμό φυσικά είναι ακρογωνιαίος λήθος της στρατηγικής αυτής. Πρόθεση των δεσμεύσεών μας, συνεργασία με διεθνείς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα με τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, το σχέδιο σχεδίου δράσης εντοπίζει κάποιους τομείς συμπληρωματικότητας, συντονισμού για εξασφάλιση της συνοχής, για την ενίσχυση του συντονισμού και για την διεύρυνση της συνεργασίας. Τρίτον, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση των δυνατοτήτων μας και την ενίσχυση των ικανοτήτων μας αξιοποιώντας τα διδάγματα του παρελθόντος, όπως την ομάδα επαφής για την καταπολέμηση της πειρατείας στις ακτές της Σομαλίας ή τις κρίσιμες, ε, το πρόγραμμα για τις κρίσιμες θαλάσσιες ε, λεωφόρους και τις θαλάσσιες διαδρομές. Ε, παραλαμβάνω ότι προσβλέπουμε στην άμεση έγκριση του σχεδίου δράσης προκειμένου να περάσουμε στη φάση εφαρμογής. Και φυσικά με την τυπική έγκριση δεν φτάνουμε στο τέλος της πορείας μας. Αυτό που προέχει είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του σχέδιου δράσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρόη. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη της ομάδας. Πρώτα η κυρία Άννα Γκόμες, που είναι και η συγγετριά μας για το θέμα αυτό της στρατηγικής ασφάλειας για την, εσωτερική, για την αυσιπλοεία. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Γκόμες. Thank you. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρουσιάσεις σας και για τόσα έχετε επιτελέσει όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης. Όπως είπατε είναι κάτι το ζωντανό. Ε, πρέπει να την πρόκληση του ακριβώς ε, δόθηκε αυτή η όθηση από την ελληνική προεδρία και ότι συνεχίζει τώρα αυτή την πορεία η Ιταλική Προεδρία και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να, να εγκριθεί. ότι θα γίνει αυτή η έγκριση το Δεκέμβριο, αλλά τόσο τη διαφορά την έκανε η Ελληνική Προεδρία. Τώρα έχουμε την Ιταλική και έχουμε στα χέρια μας τώρα αυτό το έγγραφο ε, αυτό το πρόγραμμα δράσης που είναι πάρα πολύ αξιόλογο και συμφωνώ με τις δράσεις που επισημαίνεται τις προτεραιότητες και βλέπουμε αυτά μας που ασχολούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποτυπώνονται και να καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα δράσης. Πάρα πολλά εξαρτώνται από την πολιτική βούληση, όπως είπε η κυρία η κυρία Γκμίντερ. Αυτό θα να δούμε. Τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, πού μπορούμε ε, να βοηθήσουμε και να δώσουμε καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να κινηθούν. Και εμείς πρόθυμα θα ανταποκριθούμε σε αυτά που ζητείτε. Πάρα πολύ αρέσουν η... αυτό το οποίο λέτε για περισσότερη συνεργασία ε, στρατιωτικών με πολιτικούς ε, για τις δράσεις. Και ερωτώ πρώτα απ' κύριε Ρόη, εσείς ξέρετε. Τι λείπει. Ξέρουμε τι καλύπτει αυτή η στρατηγική. Αλλά βοηθήστε μας να καταλάβουμε τι θα έπρεπε να, άλλο να καλύπτει που δεν αναφέρεται και για ποιο λόγο δεν το καλύπτεται. Μια άλλη ερώτηση. είναι ένας τομέας όπου νομίζω το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και να βοηθήσει αυτό το πρόγραμμα που έχετε αναπτύξει. Το πώς δηλαδή θα προσέξουμε τις δράσεις που έχουν σχέση και με ιστορική και εξωτερική ασφάλεια, φερειπίν κάποιες επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ε, ε, ενωσιακές αλλά είναι όπως το τρίτον μετά το Μαρινόστρομ αυτή τη δράση που ανέλαβε η Ιταλία ξέρω ότι δεν είναι τώρα θέμα μετανάστευσης και συνοριακού ελέγχου έχουν τους, τη λαθρομετανάστευση έχουμε την εμπορία ανθρώπων αλλά μια τέτοια πρωτοβουλία και εγώ ήμουν μεταξύ αυτών που ήθελα να δοθεί μια όθηση σε αυτή την ευρωπαϊκή ε, πρωτοβουλία, να υπάρξει υποστήριξη προς την Ιταλία και η οικονομική, να γίνει επομένως καθεαυτού ευρωπαϊκή επιχείρηση αυτή, πέραν του θέματος μετανάστευσης. Να έχουμε δηλαδή και στοιχεία και στόχους σχετικούς με την ασφάλεια. Γιατί είδατε τώρα τι έγινε με το Ισλαμικό κράτος που δράσει στην Λιβύη. Βρίσκονται δηλαδή λίγες ώρες μακριά από τις ευρωπαϊκές ακτές. Άρα να καλύψουμε περισσότερα, περισσότερους τομείς και όχι μόνο τη μετανάστευση. Να καλύψουμε και τα θέματα ασφάλειας. Δεν συμφωνείτε ότι έτσι θα μπορούσε να είναι ε, μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να χρηματοδοτηθεί από την Ευρώπη και έτσι να έχουμε όλες τις συνέργειες που πρέπει. Και βεβαίως και μιλάμε για μια θαλάσσια λεφόρ πάρα πολύ σημαντική. Ακριβώς όπως αναφέρατε κι εσείς. Επίσης, μήπως μπορείτε αν όχι τώρα εν ευθέτω χρόνο να μας ε, δώσετε κάποια άλλα στοιχεία για κάποιο είδους ε, περιστατικά που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στον κόλπο της Γουινέας. Γιατί όλα αυτά τα οποία γίνονται έχουν υπόψη μας ότι υπάρχει εκεί πειρατεία όπως και στις ακτές της Σομαλίας. Είναι γεγονό ότι στο, στον κόλπο τη Γουινέα έγινε κάτι τέτοιο, αλλά αργότερα προέκυψε από αυτό που μάθαμε ότι έχουμε τέτοια πολλά περιστατικά πειρατεία για τα οποία κανεί δεν μιλά. Έχουμε λαθρεμπόριο πετρελαίου στην Ιγυρία επίσης. Εκεί όπου είναι συνένοχοι και ευρωπαϊκές εταιρείες στο σαν τομέα και πριν σε μικρή νησιωτική χώρα, εκεί έπρεπε να, ε, να, υπάρξει ε, επέμβαση για δύο σκάφη, για δύο πλοία, τα οποία κάναν λαθρεμπόριο πετρελαίου. Ήταν εμπλεγμένη εκεί μια σουηδική εταιρεία. Φτωχό το κράτος αυτό, ούτε να δεν είχε λεφτά να δικάσει τους συλληφθέντες. Επίσης έχουμε και ε, κάποιον ε, κάποιον σχολταν με ναυλώσεις πλοίων από τη Μάλτα και τώρα έχουν παραπεμφθεί σε διαιτησία για την οποία κάνουν δεν έχουν τα χρήματα οι εμπλεκόμενοι και θα πρέπει να βοηθήσουν αυτές τις χώρες. Είναι χώρες ΑΚΕ γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, είμαι σίγουρη, εκτός από αυτές που ξέρω. Άρα, μήπως μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι γίνεται από πλευράς πειρατείας και, και, και άλλων ε, ε, εγκλημάτων στον κόλπο της Γουινέας. Είναι θέματα ασφάλειας, θαλάσσης. Επίσης, βλέπω, λέτε για τη δράση 1, 3, 2 και 1, 3, 3 που λέει κάτι για λαθρεμπορία, για μεταφορά λαθρομεταναστών. Τι μπορεί να γίνει εδώ. I'd like to say that Και ε, τι θα μπορούσε να γίνει άμεσα για, ε, όσον αφορά αυτές τις δράσεις. Δράση 5. Κυρία Μογκερίνη, βεβαίως και ήδη έχει κάνει τη διαφορά. Είδαμε τι έγινε στο Συμβούλιο Υπουργών ε, Αμήνης. Πήγε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Είδαμε τι στο Twitter. Είπε τα πράγματα ξεκάθαρα, να τα ακούσουν όλοι όπως θα έπρεπε να γίνει. Και Θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει ο συντονισμός που χρειάζεται μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε, τον, ε, έχουμε την κυρία Μαγκυρίνη που είναι και αντιπρόεδρος και εκτός από το, την επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και όπως υπάρχει στο στρατηγικό τμήμα υπάρχει στον πολιτικό μια δύναμη ταχείας απόκρισης μεταλλευτούμε τις δυνατότητες των κρατών μελών να εμπλακούν οι υπηρεσίες η ΕΣΕ, το Γαλιλαίος, το Κοπέρνικος ό,τι έχουμε ή τη Frontex, την εξωτερική την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, Europol και Βεβαίω δεν μπορώ παρά να σας ε, να συμφωνήσω, να σας υποστηρίζω σε αυτό το οποίο λέτε. Όπως είπε η Γκίντερ, για την συνεργασία, για κοινή κατάρτιση, εκπαίδευση, απόκριση δεξιοτήτων, για την ε, ακτοφυλακή αυτό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό. Αλλά να γίνει θα χρειαστεί πίεση και θα πρέπει αυτό να αναγορευτεί σε προτεραιότητα. Κάποιοι που έχουν τις πληροφορίες, που ξέρουν και θα μας βοηθήσουν. Και έτσι να έχουμε την ενημέρωση για τις πληροφορίες που έχει ο καθένας Οπότε και με τη συνεργασία θα καταστεί προφανές ποια είναι τα πλέον εκτήματα. Άρα εδώ χρειάζεται πρωτοπορία και ηγεσία και πρωτοβουλία ενωσιακή και ευρωπαϊκή. Τέλος, να σας τονίσω ότι θα προσφέρει ενδιαφέρον όπως είπαμε πριν για, την, για τον κόλπο της Γουινέας και την πειρατεία, να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους, τις σημαντικές ε, θαλάσσιες λεωφόρους. Χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση, να υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε, να ενημερωθούμε. Θα μπορούσαμε αυτούς που χρησιμοποιούν τις, ε, τις λεωφόρους να τους φέρουμε εδώ να μας τα πούν. Γιατί έχω επίσης ε, κάνει κάποια έκθεση για το CBRN. Για χημικά, βιολογικά κλπ. Όλοι μιλούμε για αεροδρόμια, αλλά δεν κάνουμε αρκετά και για τα λιμάνια όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά τους σχετικούς κινδύνους για τις απειλές αυτές που είπαμε για το CBRN χημικά κλπ. για τη διασύνδεση ε, και ξαναλέω προσοχή γιατί το χαλιφάτο βρά ήδη στην Λιβύα υπάρχει κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων Όλοι λέμε πω πω ότι απειλές έχουμε από τους μετανάστες. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι μετανάστες αποτελούν απειλή. Αλλά έχουμε και τις αληθεί απειλές, τις άλλες απειλές, τις οποίες δεν τις προσέχουμε αρκετά κατά τη γνώμη μου. Και αυτό επομένως το κάνουμε προτεραιότητα. Τέλος. Έχουμε τη δράση 5-2-2 για, σε σχέση με το ορίζον 2020 και θα πρέπει να υπάρξει προοικοδότηση και το ορίζον 2020 τώρα ε, προβλέπει την διπλή χρήση αλληλική πολιτική. Με σίγουρος ότι καλύπτεται. Οπότε αυτό το εκμεταλλευτούμε. Και, και εδώ χρειάζεται όμως ε, ηγετικό πνεύμα, ηγετική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν τραγικό το τι έγινε στι τελευταίε χώρε, είπε η κυρία Μπεριάλε και για την Πορτογαλία, σε πολλέ ναυτικέ χώρε, α το πούμε. Είχαμε την κρίση, είχαμε αυτά τα ηλίθια μέτρα ε, τα οποία ελήφθησαν κατά της κρίσης, οπότε και είχαμε περικοπή πολλών μας δυνατοτήτων και στον ε, στρατιώτη στον πολιτικό τομέα, αλλά και για τη θάλασσα. Και έτσι κολοβόθηκε και η μακρόπνοη ε, θαλάσσια πολιτική μας και η βιομηχανία, ναυπηγεία. Άλλα λέγαμε και άλλα κάναμε τελικά. Να, πού που χρειάζεται επομένω πρωτοβουλία, ηγετική στάση από την ε, πάτη εκπρόσωπο, την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω την Τελική Προεδρία. Έχει επίγνωση του τι χρειάζεται και τι διακυβεύεται. Σας ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Θα ήθελα να συμφωνήσω με μια ερώτησή σας. Και να το απευθύνω και στα τρία μέλη του πάνελ. Τι λείπει από αυτό το σχέδιο δράσης είναι αρκετά εκτεταμένο για να αντιμετωπίσει το εξαρτικά δυναμικό περιβάλλον θαλάσσιας ασφάλειας ε, σε όλες σχεδόν τις θάλασσές μας. Είτε στη Βαλτική, είτε στη Μεσόγειο, είτε στη Μαύρη Θάλασσα, στις ακτές της Αφρικής, στην Ανατολική Ασία. Τι γίνεται με, το εξωτερικό, με την εξωτερική πτυχή του σχεδίου δράσης. Πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο σας ερώτημα. Τι μπορεί να προσθεθεί. Και στην γεωγραφική πτυχή. Αποφασίσαμε εγώ και οι συνάδελφοι οι διπλωμάτες να να σκεφτόμαστε έτσι παγκόσμια και να δρούμε τοπικά. Ε, είναι ισορροπημένο το σχέδιο δράσης γιατί πρέπει πράγματι να υπάρξει μια ανάλυση. Να πω λίγο κάτι για την πειρατεία στον κόλπο της Γουινέας. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς πειρατεία αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας είναι ληστεία εν πλώ. Δηλαδή ε, λαμβάνει χώρα σε μια περιοχή που είναι υπό την δικαιοδοσία ενός ε, παράκτιου κράτους. Και επίσης δεν αναφέρονται τα περιστατικά όλα σύμφωνα με την γνώμη του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Δεν αναφέρονται όταν είναι σε κάποια χωρικά ύδατα. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ανώνυμη γραμμή για να καταγγέλλονται. Αλλά κατά την άποψή μου αντιμετωπίζουμε διεθνές οργανωμένο έγκλημα που έχει εξελιχθεί. Ξεκίνησαν με απλά έτσι πράγματα, με απλή ένοπλη ληστεία και έφτασαν σε αυτά τα οποία περιγράφει η κυρία Γκόμες. Ε, και έχουν προχωρήσει και στο πετρέλαιο, κάτι το οποίο βεβαίως είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ο κύριος Ρόι, γιατί κάποια από αυτά τα ζητήματα αφορούν και εσάς. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με τα πυρηνικά, βιολογικά, βιολογικά όπλα κτλ. Υπάρχει ήδη μια πρωτοβουλία από το 2010 που λέγεται Κέντρα Αριστείας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πράγματι λύνουμε και αντιμετωπίζουμε και μια ανάγκη. Ίσως πρέπει να δούμε καλύτερα πώς μπορεί να καλύψουμε το θέμα αυτό και στον τομέα της ε, θαλάσσιας ασφαλείας. Και το αναφέρεται. Το τι δεν ε, περιέχεται τώρα. Ε, εγώ θα έλεγα από την εξωτερική πτυχή είμαστε ικανοποιημένοι. Και υπάρχουν κάποια ζητήματα που ίσως να μην αναφέρονταν στην στρατηγική ασφάλειας αλλά υπήρχαν στο κοινό ανακοινωθέν π.χ. το ζήτημα έρευνας και διάσωσης ε, και εγώ θα το βλέπα και αλλιώ. Υπήρχε κάτι το οποίο αναφέρθηκε στην κοινή μας ανακοίνωση και αφορούσε τους ε, ιδιώτες ε, ενόπλους ε, προσωπικό ασφαλείας. Αλλά συνολικά θα έλεγα ότι το βλέπουμε θετικά και ξεκίνησα λέγοντας πως δεν είναι τελείως αυτό το κείμενο δεν εξαντλεί το θέμα είναι το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι θετικό οπωσδήποτε και υπάρχει οπωσδήποτε περιθώριο να ε, εξελιχθεί. Για το ζήτημα του κόλπου της Γουινέας έχω λίγα να προσθέσεις. Να προσθέσω. Οπότε οι συναδελφοί μας θα έρθουν να παρουσιάσουν ε, και τη στρατηγική του κόλπου του Γενέας μαζί με το υπόλοιπο ε, σχέδιο δράσης. Για την ε, στρατηγική, την συνεργασία τη στρατιωτική με το πολιτικό προσωπικό αναφέρθηκε, εσωτερική εξωτερική πτυχή επίσης για τις επιχειρήσεις η επιχείρηση τρίτων ε, μόλις ξεκίνησε και νομίζω πως ε, ο διευθυντής ε, της Frontex είπε πως είναι μια επιχείρηση περιπολιών στη θάλασσα, παρακτίων κτλ. Αλλά οπωσδήποτε και η διάσωση είναι πρώτη προτεραιότητα. Οπότε υπάρχει ήδη μια τέτοια πτυχή. Τέλος, για τον ρόλο και τη βοήθεια του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας, ε, οπωσδήποτε συνεχίζουμε να βασιζόμαστε επάνω σας ε, και Ευχαριστώ ε, να τα ξαναπούμε και η πρόσκληση βεβαίως και σε εσά εννοείται. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκμίντερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους, τον κύριο Ρόι και την κυρία Ιμπεριάλε. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι Ποια η κοινή θέση, αν υπάρχει κοινή θέση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην αυσιπλοεία και σε σχέση με αυτά που αναφέρονται και στο Διεθνό Οργανισμό Ναυτιλία. Εμεί είμαστε υπέρ ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέρ τη κοινή θέση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλία, ώστε να έχουμε περισσότερη διαπραγματευτική ισχύ όταν μιλούμε για τι διεθνεί προδιαγραφέ. Δυστυχώ δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη σε μια ενιαία θέση. Οπότε δεν ευωδόθηκε αυτή η πρόταση της κοινή προσέγγισης που είχαμε υποβάλει και πραγματικά είναι κρίμα που δεν τελεσφόρησε αυτή η πρωτοβουλία. Πάντως ευχαριστώ την ε, Ιταλική Προεδρία γιατί προσπάθησε για πολύ καιρό να προωθήσει αυτή την πρόταση που δυστυχώς όμως να βάγισε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να επανέλθουμε. Για τα υπόλοιπα δεν έχουμε πρόβλημα, είμαστε ικανοποιημένοι, θεωρούμε ότι είναι πλήρες το σχέδιο δράσης. Αναφερθήκατε βέβαια και στο εθνικό επίπεδο. Μερικές δράσει του σχεδίου δράσης γίνονται μόνο σε εθνικό επίπεδο και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί όλα ξεκινούν σε τελική ανάλυση από τα κράτη-μέλη. Γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Εμεί θα διευκολύνουμε, θα παρενέσουμε, θα προωθήσουμε θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση, αλλά είναι σημαντικό τα ίδια τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη στρατηγική στην πράξη και εμεί θα αξιοποιήσουμε τι δικέ του προσπάθειες για να επιφέρουμε μια προστιθέμενη αξία. Για τον ορίζοντα 2020 εξετάστηκε εκτενώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είπαμε τη χρήση να χρησιμοποιηθεί μόνο στις πολιτικές εφαρμογές. Νομική βάση πάντως υπάρχει, υπάρχουν δυνατότητες και βρήκαμε και μια καλή διατύπωση, μια εύστοχη διατύπωση και στο σχέδιο δράσης και χαιρόμαστε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Έχω και μια επιπλέον ερώτηση, κυρία Κμίντερ, μετά τα τελευταία σας σχόλια. Προς εσάς και προς τους υπόλοιπους καλεσμένους, για τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας συγκεκριμένα και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Από ό,τι ξέρω, θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Υπάρχει πρόοδος ε, που βρισκόμαστε ακριβώς. Δεν είμαι η Δήμονα ε, για θέματα Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Δεν ξέρω, εσείς Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Πάντως, τα κράτη-μέλη είναι μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθεστώς παρατηρητή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε βέβαια κάποιες συντονιστικές προπαρασκευαστικές ε, συνεδριάσεις προκειμένου να συντονίσουμε τις θέσεις μας και να συνεννοηθούμε πριν τις συνεδριάσεις. Αυτό μερικές φορές ε, μας βγαίνει, άλλες φορές δεν ε, καταλήγουμε σε κοινή θέση. Πάντως δεν έχουμε αυτόνομη έδρα όπως σε άλλες περιφερειακές οργανώσεις εκεί που μιλούμε για εμπορικά θέματα ή αλληλευτικά εκεί υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για επιμερισμένη αρμοδιότητα και μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας είναι τα κράτη-μέλη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια. Η κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ. Δύο-τρία σχόλια. Ορίζον 2020. Χαίρομαι που είπατε ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και μια και η Γερμανία προχωρεί ολοταχώς και μάλιστα μέχρι και όπλα προς τους Κούρδους ε, χορηγεί. Ελπίζουμε με κατάλληλη να αλλάξει η κατάσταση. Άκουσα και ίσως θα μπορέσουμε να προσκαλέσουμε έναν ε, ε, εμπειρογνώμονα της Chatham House, γιατί έχουν ε, καταρτήσει μελέτη για τα αποτελέσματα της πειρατείας ή της ένοπλης ληστείας στον κόλπο της Γουινέας. Θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να καλέσουμε κάποιον εμπειρογνώμονα από, το, αυτούς για να μας παρουσιάσουν ή να μας ενημερώσουν πιο διεξοδικά για τα θέματα αυτά της πειρατείας στον κόλπο της Νέας Γουινέας. Για το CBRN, τις απειλές χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών μέσων. Εμείς προσπαθούμε να, συνεργαστούμε με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που είναι καθήλια αρμόδια για τα θέματα CBRN αλλά όπως βλέπετε υπάρχει αλληλεπίδραση της εσωτερικής με την εξωτερική διάσταση. Θα μπορούσαμε λοιπόν από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να οργανώσουμε μια πρωτοβουλία και να καλέσουμε εμπειρογνώμονες ώστε να αντιληφθούν και τα κράτη-μέλη ότι τους παρακολουθούμε για τα θέματα αυτά. Τώρα, για το ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας ε, που είναι και ένοπλο. Δεν ανησυχούμε μόνο για την αυσιπλοεία. Βέβαια, σε θέματα ναυτιλίας η κατάσταση είναι πιο πιεστική και πιο ανησυχητική. Και πραγματικά μας προβληματίζει και μας ανησυχεί ότι παραλείπεται αυτό το θέμα. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν να το θέσουμε προς συζήτηση σχετικά σύντομα και να ζητήσουμε και πάλι από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσουν για την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριος Δρογεύσκη. Κύριε Πρόεδρε, έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Για το σύστημα, για το πρόγραμμα Κοπέρνικο. Σε ποιο βαθμό μπορεί το Κοπέρνικο να βελτιώσει τις ε, δραστηριότητες ε, και τις επιχειρήσεις αυτής της ε, στρατηγικής. Βέβαια είναι μια πιο μακροπρόθεσμη η προοπτική του Κοπέρνικου, αλλά με ενδιαφέρει σε ποιο βαθμό μπορεί η ανάπτυξη αυτού του συστήματος να διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής για την ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία για τα έγγραφα, αλλά και για τη συνεργασία με την Τουρκία, ποιες είναι οι προοπτικές ε, περαιτέρω συνεργασίες με την Τουρκία, γιατί νομίζω ότι και για την ανατολική διάσταση η συνεργασία αυτή έχει μεγάλη σημασία. Σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας, σε κάποιον συγκεκριμένο. Όχι, νομίζω ότι είναι προς όλους ε, αυτέ αυτές οι ερωτήσεις. Ωραία, παρακαλώ λοιπόν τους καλεσμένους μας να δώσουν απαντήσεις. Ξεκινήσουμε από την ε, κυρία Εμπεριάλε, μετά τον κύριο Ρόι και τέλος την κυρία Κμίντερ. Εκτός μικροφώνου κυρία Εμπεριάλα. Done the utmost to put... Έκανα ό,τι μπορούσα τόσο ώστε να χρησιμοποιήσουμε το Κοπέρνικο ή και τα άλλα προγράμματα. Όλα εκείνα τα οποία λίγο πολύ αφορούν την καταθάλασσα ασφάλεια και να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή. Όπως είπαμε, όμως, ε, ακόμα είμαστε στην αρχή της διαδρομής, δεν την έχουμε ολοκληρώσει. Και να δούμε αν ε, αυτό το παιδί, αυτό το μωρό μεγαλώσει που αυτό το πρόγραμμα δράσης και ενηλικιωθεί. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Στην αρχή του έργου. Και θα πρέπει να δοθεί μια όθηση στην επόμενη Προεδρία προεδρίες θα έλεγα, γιατί δεν πρόκειται για κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε έξι μήνες, μια που θέλουμε διαφορετικούς τομείς να ε, κάνουμε να προοδεύσουν. Κύριε Ρόι, έχετε λόγο. Thank you. Σας ευχαριστώ για τον Κοπέρνικο. Δεν είμαι ειδικό, αλλά Οπωσδήποτε. Θα πρέπει να ενημερωθούμε. Και σε σχέση με το πρόγραμμα δράση για την καταθάλασσα ασφάλεια, βεβαίως και μας δίνει δυνατότητες το πρόγραμμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την θάλασσια ασφάλεια. Και να δούμε πώς με τον καλύτερο τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το πρόγραμμα. Είναι θέμα του πώς θα το υλοποιήσουμε για την Τουρκία. υπάρχει κάποιος διάλογος και συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Και αρμόδια είναι η Επιτροπή Κοινή Πρωτοβουλία. Εμπλέκονται τα κρατη ούτως ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ότι έχει συμφωνηθεί. Ούτε εδώ είμαι ειδικό βέβαια. και έχουμε και επίσης και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για τον Κοπέρνικο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε μια συγκεκριμένη δέσμη για τον Κοπέρνικο, για συλλογή και διάδοση πληροφοριών. Τώρα κοιτάμε να δούμε ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουμε, ποια δεδομένα μας ενδιαφέρουν από τον Κοπέρνικο, αλλά σύμφωνα με την τελευταία πληροφορία μου είναι πως βρισκόμαστε ακόμα στην φάση την ενιολογική. Αλλά καθώς, ε, εννοώ βεβαίως ε, του σχεδιασμού, αλλά καθώς βεβαίως δεν είμαστε, δεν το ασχολούμαι εγώ καθημερινά, δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Τώρα για την Τουρκία και τον διάλογο για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τις θαλάσσιες μεταφορές ε, μιλάμε τακτικά, είμαστε σε επαφή και εγώ έχω πάει στην Τουρκία και για να τους εξηγήσω το θέμα αυτό υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Πλησιάζουμε το τέλος της συνεδρίασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. για την θαλάσσια στρατηγική ασφαλείας. Να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Γκόμες, την εισηγήτρια, για την επαγγελματική της ε, παρέμβαση και συνεισφορά και τους και τις ε, βουλευτές ειδικά τη ε, μέλη της υποεπιτροπής μας λύεται η συνεδρίαση η επόμενη συνεδρίαση 3 Δεκεμβρίου ευχαριστώ